Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Καλησπέρα σα ε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μα δύο σχεδόν θαμώνε τη Επιτροπή μα. Εντάξει, για τον ε, Πτέραρχο δεν ισχύει αυτό ακόμη, αλλά ω προ τη θέση του και την ιδιότητά του ως ανώτατου διοικητή της συμμαχικής ε, διοίκησης μετασχηματισμού και με τον προχατοχό σας ε, είχαμε πολύ συχνές συναντήσεις και μαζί με την κυρία Αρνού, την Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο τακτικές συναντήσεις και κρίναμε σκόπιμο και ενδιαφέρον να ανανεώσουμε αυτή την επικοινωνία μας, γιατί η συζήτηση για τις στρατικές δυνατότητες εξακολουθεί να είναι πολύ έντονη και σφοδρή και στο ΝΑΤΟ και αύριο θα έχετε τη διπογική διάσκεψη του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε την άμυνα ε, ως ε, σημείο του της ημερήσιας διάταξης ε, της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου. Οπότε και για το θέμα αυτό δημιουργούνται αρκετές προσδοκίες, γι' αυτό και παρακολουθούμε με ιδιαίτερα ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Και χθε μάλιστα πολύ πρόσφατα είχαμε ε, επίσκεψη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και είδαμε διεισόμαση τις προσπάθειες που γίνονται για διάφορα θέματα και ο Παλωμέρος ε, πολύ συχνά το τελευταίο καιρό σε διάφορα φόρα τόνισε τη συνέργεια που υπάρχει μεταξύ του οργανισμού και του ΝΑΤΟ, τη έξυπνης άμυνας και του pooling and sharing, της συνένωσης δηλαδή και κοινής χρήσης των πόρων. Και ελπίζω ε, μετά την εξοικείωσή μας με τους ε, όρους να εξοικειωθούμε και με την ε, έμπρακτη εφαρμογή τους. Να περάσουμε λοιπόν από τα λόγια στα έργα και σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο Κορυφή του Δεκεμβρίου, σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε δημόσια ακρόαση με εκπροσώπους βιομηχανίας και με τον Γάλλο Υπουργό Άμυνα πριν από δύο εβδομάδες. Και παρόλα αυτά πλανάται κάποιος σκεπτικισμός, ακόμη και μεταξύ μας. Και δεν βλέπουμε και πολύ συγκεκριμένες και αυτές προτάσεις επί το παρόντος. Οπότε από τις συζητήσεις μια διαπίστωση που είναι κοινή είναι ότι έχουμε κυρίως από τα θέματα της στρατικών ικανότητων τα πιο, τις πιο μεγάλες προσδοκίες και εκεί μπορούμε να αναπτύξουμε κάποια κοινά προγράμματα που καλό θα ήταν να, να ε, αναφερθούν και από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να μην περάσουν απαρατήρητα και ελπίζουμε να φανεί τέτοιο ενδιαφέρον από τη Σύνοδο Κορυφής. Μιλούμε για, την για τον εναέριο ενεφοδιασμό, ε, επίσης το θέμα των ντρόν, αυτών των μη επαδρομένων αεροσκαφών και ήταν ατυχής οι λύσεις που αναγκάστηκαν να θετήσουν μερικέ χώρε, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και πόσο σκόπιμο και επίκαιρο είναι να τα θέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι λοιπόν μερικά από τα θέματα που μας απασχολούν, που βρίσκονται επιτάπητος και θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από την κυρία Αρνού να κάνει την πρώτη παρουσίαση. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πτέραρχο Παλωμερός και θα ακολουθήσει η συζήτηση η κυρία Αρνού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ επ' ευκαιρία και για την επίσκεψη που πραγματοποίησε η Επιτροπή σας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα ε, τον ΕΝΤΑ. Είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος αυτός για μα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ικανοτήτων, ε, φυσικά είναι μεγάλο προνόμιο που έρχομαι εδώ, ε, όχι για πρώτη φορά με τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, τη συμμαχική διοίκηση μετασχηματισμού, αλλά ιδιαίτερα με τον πτέραρχο Παλομερό. Αυτό είναι αυτή η απόδειξη τη στενή συνεργασία που έχουμε με το ΝΑΤΟ. Και ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της ε, Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ για τα θέματα των ε, ικανοτήτων, ικανοτήτων. Να αναφερθώ σε κάποιε ίσως ε, και σε κάποιες καινοτοπίες που όλοι τις γνωρίζουμε, γιατί είχατε πρόσφατα και σχετικές δημόσιες ακροάσεις. Το υπόβαθρο είναι γνωστό, οι προκλήσεις και οι απειλές είναι αμή άλλο πολυάριθμες και σημαντικές Οπότε το κόστος αντίδρασης ε, στις ε, προκλήσεις αυτές αυξάνεται με γεωμετρικό τρόπο γιατί και στις αρχικές επενδύσεις αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων ε, είναι τεράστιες οι δαπάνες που απαιτούνται. Δεν μπορούμε λοιπόν να διακινδυνεύσουμε τι ζωές ε, είτε στρατιωτών μας ή άμαχου πληθυσμού. Και από αυτή την άποψη οι υπολογισμοί των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υφίστανται περικοπές ε, και μερικές φορές και η άμυνα υπόκειται σε αυτή την δημοσιονομική λιτότητα. Πολύ περισσότερο μερικές φορές και από άλλου Και όταν αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τα δημοσιονομικά θέματα Νομίζω ότι το πρώτο ζητούμενο στη συζήτηση είναι να τηρήσουμε τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις και να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα και άρα να περικόψουμε κάπως τον προϋπολογισμό. Οπότε ξεκινούμε από το σενάριο, από την υπόθεση ότι και ο προϋπολογισμός για την άμυνα θα περικοπεί. Χρειάζομαστε όμως ε, κάποιες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις που θα αναγνωρίζουν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην άμυνα και ανάγκη μεγιστοποίησης ε, και βελτιστοποίησης της προσπάθειας που κάνουμε σε αυτές τις ε, δύσκολες συνθήκες και τους χαλεπούς καιρούς. Επίσης, πολύ συχνά εξετάζεται την εξάρτηση που έχουμε μερικές φορές ε, κατά 80% από τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τις πρόσφατες επιχειρήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν κατά 80% σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη κάποιων στρατιωτικών ικανοτήτων. Και το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν σαφές πια και ξεκάθαρο και αυτό θα το σχολιάσει πολύ καλύτερα από μένα ο πτέραρχος Παλωμέρος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δήλωσαν δεν θα συνεχίσουν συστηματικά να παρέχουν το 80% των στρατιωτικών ικανοτήτων ε, και είπαν κάντε ό,τι μπορείτε και μόνοι σα από εδώ και πέρα. Οπότε αντιμετωπίζουμε αυτή τη δυσκολία και έχουμε αυτή την προοπτική πια ότι στα τέλη του έτους, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής τους ε, έχουν στο πρόγραμμα και το ζήτημα της άμυνας. Αυτό που ίσως αναμένεται και τουλάχιστον ε, εμείς ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε, δεδομένη τη ανάγκη και τη κατάσταση να δοθεί προτεραιότητα στην ε, άμυνα, γιατί το θέμα της ασφάλειας είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους, αλλά είναι σημαντική προτεραιότητα που θα δοθεί στην άμυνα, που πρέπει να δοθεί στην άμυνα και γι' αυτό και βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφή στο πρόγραμμα. Ε, η άμυνα είναι ένα σημαντικό παράγοντα κοινοτομία και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Υπάρχει λοιπόν το θέμα τη ασφάλεια, αλλά και το θέμα το, το οικονομικό. Δημιουργείται με την άμυνα μια τεχνολογική βάση στην αμυντική βιομηχανία και πολλέ θέσει απασχόληση. Οπότε με την προτεραιότητα τη Άμυνα θα πρέπει ταυτόχρονα να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μα με τη συνεργασία ή με την ενίσχυση τη συνεργασία και του συντονισμού μα. και επίση να δώσουμε προτεραιότητα και στη μελλοντική μα προετοιμασία και στον εξοπλισμό αλλά και στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Γιατί πολύ συχνά εκεί γίνονται οι μεγαλύτερε θυσίε όταν γίνονται δημοσιονομικέ περικοπέ και ιδιαίτερα στο θέμα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης μπορούμε να κάνουμε μια σαφή εράρχηση των προτεραιοτήτων μας που είναι ε, απαραίτητες και από στρατηγική άποψη και για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και επίσης για να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές συνέργειες ώστε οι κοινοτικές πολιτικές και η ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, να μην ε, δεξαγάγονται παράλληλα. Θέλουμε μια ολιστική προσέγγιση, σφαιρική προσέγγιση από όλε τι ε, ενωσιακέ πολιτικές. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους διάφορους μηχανισμούς και τα εργαλεία που έχουμε ώστε να κάνουμε διτή χρήση των ε, μέσων μας. Οπότε ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα συμβάλλουμε στην προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής μέσω της έκθεσης της Καθιάστων και των εργασιών των Υπουργών Άμυνας ε, θα υποβάλουμε πολύ ρεαλιστικές προτάσεις και θα προσπαθήσουμε να επισήσουμε την προσοχή των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε σημαντικά προγράμματα που έχουν κεφαλαιόδη σημασία από στρατιωτική άποψη. Για παράδειγμα το θέμα της, του, ενα, του ανεφοδιασμού στον αέρα ε, που είναι πολύ σημαντικό θέμα και εκεί αναμένεται πραγματικά μια ευρωπαϊκή απόκριση, γιατί στο Σικάγο η αρχική κρατών κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ περιμένουν μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον αέριο εφοδιασμό σε καύσιμα. Επίση, ό,τι αφορά τους δορυφόρου επικοινωνία τηλεπικοινωνιών και αυτό το θέμα, οι δυνατότητε μα και οι ικανότητέ μα σε αυτό το επίπεδο είναι σημαντικέ. Επίση θα πρέπει, και συμφώνησα γι' αυτό η Υπουργή Άμυνα, να εντοπίσουμε του πρωτοπόρου τομεί που είναι η πιο σημαντική και επίσης ενδεικτική τη σύγκληση που μπορούμε να έχουμε μεταξύ των υπόλοιπων κοινοτικών πολιτικών και της πολιτικής άμυνας. Έχουμε για παράδειγμα το Remote Piloting System, τα ε, αεροσκάφη που, τα μη επανδρομένα που, τα, που εξ αποστάσεως ε, τηλε, τηλεκατευθυνόμενα κατά κάποιο τρόπο αεροσκάφη και υπάρχουν κάποια τεχνολογικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να τηρηθούν οι κανόνες που έχουν και ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τις αγορές από τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουμε και πάλι να έχουμε όσο δυνατόν ε, κοινή χρήση των πόρων είτε στη χρήση είτε στους τρόπους εφαρμογής των αγορών που έχουν γίνει, των προμηθειών που έχουν γίνει και να προετοιμάσουμε από κοινού τις επερχόμενες γενναίες. Τα συστήματα τηλεκατεύθυνσης των αεροσκαφών και των μικρών και των μεγάλων αεροπλάνων. Και μάλιστα κάτι τέτοιο έχει και δει χρήση, στρατιωτική και μη στρατιωτική. Ένα δεύτερο τομέα που έχει κεφαλαιόδη σημασία και εκεί επίση οι Υπουργοί Άμυνα για το θέμα αυτό συμφώνησαν, αφορά το θέμα της άμυνας στον κυβερνοχώρο. Βέβαια αυτή η έννοια είναι πολύ γενική, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι ζωτική σημασίας. Και είπαμε να επικεντρωθούμε και στο θέμα αυτό σε ορισμένες δράσεις για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και να δυσκετάσουμε τις ανησυχίες των κρατών μελών θα επικεντρωθούμε σε κάποιους τρόπους εξάσκησης ή κατάρτισης και στην προστασία των δικών μας ε, ικανοτήτων και αποστολών και στρατιωτικών και πολιτικών ώστε να, έχουμε, να μπορούμε να πτήσουμε και μονάδες ε, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ένα ε, άλλο σημαντικό θέμα για τη Σύνοδο Κορυφή είναι η στήριξη που θα δοθεί στην αμυντική μα βιομηχανία και στην ε, έρευνα και τεχνολογία στην αμυντική βιομηχανία. Είχατε δημόσια κρόση με του εκπροσώπου τη αμυντική βιομηχανία και το μήνυμα είναι καθαρό και απερίφραστο. Γιατί τα όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων ασφάλεια και άμυνα είναι πολύ ρευστά. Γι' αυτό και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στα πλαίσια της απασχόλησης αλλά και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και πιστεύω ότι αυτό θα απασχολήσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων γιατί χωρίς τεχνολογική βιομηχανική βάση δεν θα έχουμε στρατηγική αυτονομία και άρα δεν θα έχουμε και ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Οπότε για να έχουμε στην Ευρώπη οι ικανότητες που θα μας επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε στρατηγική αυτονομία και ε, τέτοια στρατηγική είναι απαραίτητη να λάβουμε υπόψη την αμυντική μας βιομηχανία και να τη στηρίξουμε. Επίσης, θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση, αλλά δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε στην πορεία την τεχνολογική και βιομηχανική μας βάση. Γιατί οι μεγάλες βιομηχανίες που μπορούν να έχουν δραστηριότητε διτής χρήσης, αλλά κάποια στιγμή ίσως ε, απομακρυνθούν τελείως από το στρατιωτικό τομέα. Κάτι που είναι κίνδυνος και για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και για την ε, απασχόληση, αλλά και για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού μας. Άλλωστε δεν έχουν ε, όλοι τις επιλογές που έχουν οι μεγάλες βιομηχανίες. Οπότε θα πρέπει εμείς να οδηγήσουμε σε ασφυξία τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις που ασχολούνται με την άμυνα. Πολύ συχνά οι βιομηχανίες στηρίζονται στις εξαγωγές, αλλά οι εξαγωγές πολλές φορές γίνονται με μεταφορές τεχνολογίας και μάλιστα μεταφορές τεχνολογίας σε χώρες που έχουν επενδύσει στο θέμα αυτό. Ακριβώς επειδή είμαστε σε ένα υψηλό τεχνολογικό και βιομηχανικό επίπεδο, προς το παρόν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια αυτή της μεταφοράς τεχνολογίας και εξαγωγών. Αλλά αν αύριο μειώσουμε τις επενδύσεις μας και άλλες χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και άλλες συνεχίσουν με ταχύ ρυθμό τις δικές τους επενδύσεις, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα διασφαλίσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, αλλά θα βγούμε χαμένοι σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Οπότε δεν είναι αβάσιμη απεσιοδοξία, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου και να εστιαστούμε στις δυνατότητες συνέργειας που υπάρχουν μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών και των εθνικών πολιτικών. Των πολιτικών που γίνονται σε, σε διακυβερνητικό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, αλλά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο με ε, εστίαση σε συγκεκριμένα προγράμματα. Είπαμε να μην μιλήσουμε γενικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στήριξή τους, αλλά να εφαρμόσουμε αυτή τη στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στα ντρόν, για παράδειγμα, ή στην αγορά της, ε, της προστασίας στον κυβερνοχώρο. Αλλά και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και το, δικό χαρακτήρα των, το διτό χαρακτήρα των ικανοτήτων, τον στρατιωτικό και πολιτικό δηλαδή σκέλος. Χρειαζόμαστε αυτή την ε, κοινή προσέγγιση αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την τεχνολογική και βιομηχανική μας βάση. Επίσης, έχουμε υψηλές προσδοκίες από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που με συγκεκριμένες προτάσεις υποστηρίζει αυτό το διτό τομέα, στρατιωτικό και πολιτικό, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη χρήση των κοινωτικών κοντιλίων. Γιατί αφενός ε, έχουμε τέτοιες διπλούς τομείς ή κάποιες κοινέ προτεραιότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα κατάλογο με τεχνολογίες κλειδιά, Key Enabling Technologies, Έχουμε επίσης ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και επίση εκεί έχουμε ένα κατάλογο με τεχνολογίες. Μπορούμε λοιπόν να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και να συνδυάσουμε τα διάφορα κοινοτικά εργαλεία που έχουμε με τήρηση φυσικά και σεβασμό των αμοιβαίων αρμοδιότητων μα. Και λαμβάνοντα υπόψη το διτό χαρακτήρα αυτών των ικανοτήτων και των μηχανισμών που έχουμε. Και τέλος, να πω ότι τα κράτη-μέλη απαιτούν από εμά να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και γιατί πολλές χώρες είναι ταυτόχρονα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κόπτονται για, να, για την αποφυγή αυτών των επικαλύψεων. Θα συνεργαστούμε φυσικά με το ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό. Εμεί ως Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα έχουμε άμεση συνεργασία με την Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού ε, και θέλουμε και το pooling and sharing, συνένωση και κοινή χρήση και η smart defense, έξυπνη άμυνα, να μην είναι ανταγωνιστικές έννοιες μεταξύ τους. Και είναι δύο παραδείγματα που θα τα αναφέρουμε και αργότερα στη συζήτηση. Επίσης έχουμε σχέσεις με κέντρα αριστείας των κρατών μελών που έχουν λάβει και την πιστοποίηση του ΝΑΤΟ. Αυτά τα κέντρα αριστείας για την, στο Τάλιν ή στην Ισπανία για την ε, προστασία στον κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Επίσης ε, έχουμε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ για το, το πρόγραμμα των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων, ώστε εδώ να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι ανάγκες του ΝΑΤΟ και για, τις, για τους ειδικευμένους οργανισμούς, την NCIA, γιατί μίλησα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θέλουμε ε, αυτό που κάνει η NCIA για την προστασία των, ε, των μέσων του ΝΑΤΟ να τα κάνουμε και εμείς ε, σε συνεργασία για να προστατεύσουμε τα διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τις επιφυλάξεις και το σκεπτικισμό, το συζητήσαμε και στην ετήσια διάσκεψή μας, αλλά στο θέμα των ικανοτήτων μας η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να είμαστε δραστήριοι και αποφασιστικοί. Χρειαζόμαστε φυσικά τον ενθουσιασμό και την κοινή βούληση όλων, ώστε να στηριχθούμε σε κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες που θα γίνουν σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία φυσικά με τα κράτη-μέλη, γιατί η συμβολή των κρατών μελών στη Σύνοδο Κορυφής θα είναι πολύ μεγάλη και με βάση τις ιδέες, τις προτάσεις μας ε, και τους τρόπους που θα προτείνουμε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ορισμένα θέματα όπως ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ένα αέριος αναφοδιασμό σε καύσιμα, ντρόν και ούτω καθεξής. Εκεί όπου υπάρχει συμφωνία μπορούμε ήδη να προχωρήσουμε. Αυτό θα ήταν μεγάλη επιτυχία για τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Οπότε, αν καταφέρουμε να πείσουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να τηρήσουν αλόβητε τις προσπάθειες για την άμυνα και να επικεντρωθούμε στις πιο σημαντικές τεχνολογίες και στην βέλτιστη χρήση ε, των κονδυλίων και στους εθνικούς και στους, ε, στον κοινωτικό υπολογισμό νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, είχα μιλήσει για σκεπτικισμό, όχι για απεσιοδοξία. Θα δούμε. Με το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε πέσει σε απεσιοδοξία. Ελπίζω πως όχι. Πτέραρχε. Για το ACT για τη συμμαχική δίκηση μετασχηματισμού φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα που δυσκολευόμαστε να ξεπεράσουμε ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο, αλλά πάντως όσον αφορά τις ικανότητες, τις δυνατότητες που έχουμε, νομίζω πως ε, ξεπερνιούνται τα προβλήματα. Φαντάζομαι πως θα μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ελπίζω πως δεν θα, είναι ακόμα ένα θέμα, ε, μια λαβή για απογοήτευση και σκεπτικισμό. Ελπίζω, γιατί είμαι κι εγώ αισιόδοξο ε, Ας ε, διατηρήσουμε και αισιοδοξία και απεσιοδοξία γιατί η ισορροπία των δύο θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Καταρχήν, Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτές, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου και την τιμή που αισθάνομαι να βρίσκομαι ε, σήμερα εδώ δίπλα στην ε, κυρία Γιώσφα Σαρνό και ως διοικητής μια στρατηγική διοίκηση του ΝΑΤΟ που είναι κατεστημένη στις ΗΠΑ, Ευρωπαίος και Γάλλος ε, διοικητή, αν και το στρατηγείο των επιχειρήσεων είναι εγκατεστημένο στην Ευρώπη και εκεί διοικεί ο Αμερικανός διοικητής, όπως γνωρίζετε, Πάντως η ιστορία που αυτή τη στιγμή ε, γράφεται αυτή τη στιγμή ιστορία κατά τη γνώμη μου και θα πρέπει να σα ομολογήσω πως είμαι πολύ περήφανο, διότι έτσι θα μπορέσουμε να γράψουμε μια κοινή ιστορία, αυτή είναι η αίσθηση που έχω και θα προσπαθήσω να σας δώσω και κάποια παραδείγματα στη σύντομη μου παρέμβαση. Να θυμίσω ότι σε θεσμικό επίπεδο η διάσκεψη κορυφή τη Λισαβόνα του 2010 του ΝΑΤΟ θεωρήθηκε, θεώρησε μάλλον στρατηγική φύση σε την εταιρική σχέση ανάμεσα στη Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάσκεψη κορυφή του Σικάγο πριν από ένα χρόνο περίπου επανεπαβεβαίωσε τη σημασία αυτή τη ε, ιδέα για τον ΝΑΤΟ. Τον ανήκει στην ε, Ατλαντική Συμμαχία προσφέρει σε κάθε έναν από του συμμάχους ένα μοναδικό δυναμικό, μια κληρονομιά αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, και στρατηγική σύγκληση, η αλειτουργικότητα που είναι πολύ στρατηγική για να μπορούν να ενεργούν μαζί αυτές οι δυνάμεις. Είναι μια αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Αυτή τη στιγμή 21 χώρες είναι μέλη της Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα και αγωνίζεται ώστε ο προβληματισμός σε σχέση με τις ικανότητες να ακολουθεί καταρχήν την κοινή λογική αλλά και την αίσθηση της ιστορίας ώστε πραγματικά να γίνονται συντονισμένες κινήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αφορούν τις ίδιες δυνάμεις και τους ίδιους προπολογισμού. Όντως σήμερα στο πλαίσιο της συμμαχίας είμαι Είμαι βαθύτατα πεπισμένο ότι διαγράφεται μια πραγματική προοπτική για τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποκτήσουν μέσα και για μια πολιτική ασφάλεια και κοινή αμήνη συμβατέ με το δέσμευσή του προ το ΝΑΤΟ, που θα ευνοεί μια ισότιμη κατανομή των, του βάρου ή του καθήκον, όπω θέλει κανεί να μεταφράσει το burden sharing ε, ανάμεσα στις δύο όχθες ε, της ε, Ατλαντικής Συμμαχίας. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν βρίσκω για ακόμα μια φορά την Διευθύντρια της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης γιατί πιστεύω πως πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο εργαλείο αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση θετικά το, το λέω είναι ένα εργαλείο για την οικοδόμηση του μέλλοντος των, των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ικανοτήτων και υπ, αυτήν, υπ αυτόν τον, τον τίτλο χρησιμοποιούμε κάνουμε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντονίσουμε τις κοινέ μας ε, προσπάθειες. Και είναι πολύ άριθμες. Θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε για να πάρω το λόγο, για να σας θυμίσω τι είναι η συμμαχική διοίκηση μετασχηματισμού, διότι αυτή συγείται ένας Ευρωπαίος και ηθελημένα. Η Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού στόχο έχει να προετοιμάσει τη Συμμαχία στι αυρινές προκλήσει που το αύριο βέβαια ξεκινά σήμερα, προσαρμόζοντα αυτή τη Συμμαχία στι προκλήσει και στο περιβάλλον πράγμα το οποίο απαιτεί μια στρατηγική οπτική, μια εξέλιξη των ικανοτήτων και ταυτόχρονα καλύτερη εξάσκηση τον και ε, κατάρτιση των δυνάμεών μας. Με αυτό ασχολούμαι ακριβώς, με αυτούς τους τρεις άξονες και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ο μετασχηματισμός είναι μια μόνιμη διαδικασία διαρκής, ε, όχι μόνο για τη συμμαχία, αλλά μέσα στο πλαίσιο της συμμαχίας έχει θεσμοθετηθεί μέσω της διοίκησης ε, μια διαδικασίας που είναι ίσως κάπως βαριά, αλλά που είναι πολύ συγκεκριμένη γιατί ανταποκρίνεται σε επίπεδα φιλοδοξίας που απορρέουν με τη σειρά τους από μια στρατηγική ε, έννοια και οδηγούν τελικά σε εξέλιξη των στόχων ικανοτήτων. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και σε ποιο ορίζοντα. Αυτό είναι που το ΝΑΤΟ και η Συμμαχία έχουν οικοδομήσει από τη δεκαετία του 60. Μέσα σε αυτή τη δυνατότητα οικοδόμησης ικανοτήτων εφάνει σαφώς πως το ΝΑΤΟ χρειαζόταν να επιταχύνει κάποια προγράμματα γιατί όλα αυτά παίρνουν πολύ χρόνο, είναι χρονοβόρα και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί καθώς και η αλλαγή του περιβάλλοντος ήταν τέτοιου βαθμού που έπρεπε να ανταποκριθούμε επιγόντως σε ανάγκες επιτακτικές ή και επίγουσες ε, μελλοντικά. Αυτή είναι το νόημα του Smart Defense, ε, της ευφύους άμυνας που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας ε, Ράσμουσεν που ανταποκρίνεται σε, κατά κάποιο τρόπο ή είναι η παραλληλότητα, του, της, παραλληλισμός μάλλον του pooling and sharing της, κοινής, της συγκέντρωσης και κοινή χρήσης των ικανοτήτων. Αυτή η άμυνα που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε το Smart Defense, η ευφυής άμυνα, ε, βασίζεται στην εξή απλή αρχή. Πώς μπορούμε δηλαδή να δώσουμε ένα νόημα σε μια πολυεθνική προσέγγιση εκεί όπου η φυσική τάση θα μας ε, οθούσε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες ικανοτήτων μέσα σε μια εθνική λογική, όπως ε, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, αν και υπήρξαν κάποια επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασίας στο παρελθόν. Πώς λοιπόν θα προωθήσουμε τέτοιου είδους πολυεθνική συνεργασία και πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα όθηση για να καινοτομήσουμε και να βρούμε ίσως πρωτότυπες απαντήσεις, λιγότερο δαπανηρές, πιο προσαρμοσμένες, πιο στοχοθετημένες. Αυτό είναι το νόημα της εφηούς άμυνας και του pooling and sharing. Εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει ο μετασχηματισμός και προσπαθούμε να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την πολυεθνική προσέγγιση. Εξάλλου μου έχει ανατεθεί από το Γενικό Γραμματέα ω ειδικό απεσταλμένος για να υπερασπιστώ αυτή την προσέγγιση στις διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ και μάλιστα η υποδοχή είναι πολύ ευνοϊκή εν γέννη. Σήμερα έχουμε λάβει 150 προγράμματα και σχέδια συνεργασίας υπό την ΕΦΗ Άμυνα. Ε, που όλα είναι βιώσιμα και καμιά τριανταριά έχουν ήδη ξεκινήσει στην υλοποίησή τους, βασίζονται στην βούληση ενός έθνους πλαισίου να αναθέσει την ευθύνη σε μια χώρα για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου και για τη δημιουργία μιας ομάδας ε, χωρών εθελοντών που ε, εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα. το, η δίκηση μετασχηματισμού εξασφαλίζει το, την παραπληρωματικότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στα, δύο, ανάμεσα στα έθνη που συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα. Και τώρα θα μου να στραφώ στη γλώσσα του Σέξπιρ, που είναι η δεύτερη γλώσσα του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να σας δώσω μια εικόνα για την παραπληρωματικότητα. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με στόχο το κοινό όφελο. Βεβαίω, πώ μπορεί να γίνει αυτό. Η σύντομη απάντηση μπορεί να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα με τι χώρε, για τι χώρε και σε διαβούλευση με του ενδιαφερόμενου. Πρακτικά, ο, μετασχηματισμό. ο Οργανισμό Μετασχηματισμού και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα συνεργάζονται πάρα πολύ στενά για να σχεδιάσουν το μέλλον και να βελτιώσουν το παρόν με μια ε, κοινή και ουσιαστική πτυχή την βιομηχανία. Έτσι ξεκινάμε με μια κοινή κατανόηση του μελλοντικού στρατηγικού περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων που θα χρειαστούμε. Ο οργανισμός του μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ εργάζεται για το επιχειρησιακό περιβάλλον του 2030 και για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό αυτών και το στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας σημαντικός παράγοντας για το κοινό αυτό όραμα είναι πως πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από τις τρέχουσες επιχειρήσεις, ειδικά για να βρούμε που υπάρχουν ελλείψεις στις δυνατότητές μας. Αυτό κάναμε ακριβώς παραδείγματο χάρη μετά την επιχείρηση στη Λιβύη που αποκάλυψε λήψεις σε τομείς όπως ένα αέριος ανεφοδιασμός, ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, ε, εκτίμηση κατάσταση του πεδίου τη μάχη και στρατηγικών μεταφορών. Για να βελτιωθούν λοιπόν οι παρούσες δυνατότητες μας, συντονίζουμε τις προσπάθειε μας για να χρησιμοποιήσουμε τους ε, πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε από τις ε, χώρες όσον αφορά τον αέριο ε, ανεφοδιασμό στην Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ του 2010 κάτι το οποίο αναπτύσσεται για το μέλλον υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Επίσης, η συνεργασία με τη βιομηχανία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ακριβώς γιατί ο μελλοντικό ε, μετασχηματισμός, η υπηρεσία αυτή, δεν είναι μία υπηρεσία προμηθειών. Η συνεργασία λοιπόν επιτρέπει στη βιομηχανία να έχει μια καλύτερη ιδέα, ιδέα για το ποιες είναι οι απαιτήσει μας και στην ε, στρατιωτική πλευρά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι θα μπορέσει να μας προσφέρει η βιομηχανία, πότε και με ποιο κόστος. Η συνεργασία μας λοιπόν έχει κρίσιμη σημασία για τη συνεργασία και έτσι πρέπει να λάβουμε υπόψη βεβαίω και τις ε, δημοσιονομικές πιέσεις έτσι ώστε οι στατοί μας να παραμείνουν, με, να παραμείνουν εξοπλισμένοι με αποτελεσματική τεχνολογία. Και βεβαίως ε, το πνεύμα αυτό της συνεργασίας διαπνέει και το πλαίσιο του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, παρά το ότι εκ πρώτης όψης φαίνονται ανταγωνιστικές. Θα αναφέρω έναν τομέα που έχει ήδη επιδείξει αποτελέσματα. Παράδειγμα του χάρη τα ελικόπτερα. Το σχέδιο Smart Defense του ΝΑΤΟ έχει συνεισφέρει στη μείωση του χρόνου επισκευής, ενώ το pooling and sharing έχει δημιουργήσει ένα σχολείο εκπαιδευτών και άρα ε, παρέχει την, ανθρώπινη, την πτυχή του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη τυποποίησης ε, που θα προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα της πληρωματικότητας μέσω της διτής αυτής προσέγγισης και τεχνολογιών η τυποποίηση έχει ήδη βελτιώσει τη δυνατότητα των συμμάχων να συνεργάζονται και να ξεπεράσουν τα εμπόδια μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής οργάνωση και χωρών. Θα ήθελα να επισημάνω, παραδείγματος χάρη, τους ε, κανόνες ε, αεροπλοείας για την ε, λειτουργία και συντήρηση αεροσκαβών ή επίσης τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, κάτι το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Επίσης πρέπει να αναφέρω την ανάπτυξη των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, η οποία για εμάς είναι βέβαια κάτι το πολλά υποσχόμενο. Πρέπει να υπάρξει μια νέα γενιά τέτοιων αεροσκαφών που θα είναι πιστοποιημένα για να χρησιμοποιούνται στους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Οπότε, συμπερασματικά, με συνεργασία, με διαφάνεια και με αμοιβαία εμπιστοσύνη, οι δύο υπηρεσίες μας ε, προχωρούν στην κατάρτιση τυποποιημένων απαιτήσεων με την ε, στρατιωτική εμπειρία και τις συμβουλές της βιομηχανίας. Θεωρώ πως ε, αυτή είναι η καλύτερη προστασία που μπορούμε να έχουμε απέναντι στην επανάληψη των προείδιων προσπαθειών δύο φορές. Έτσι η Smart Defense και το Pooling and Sharing, οι πρωτοβουλίε αυτές, θα μας δώσουν νέες ευκαιρίες για ε, ανάπτυξη της βιομηχανίας στο σύνολο της. Και βεβαίως ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απέτηση και ξεκινήσει ένα έργο, θα υπάρξει και το στοιχείο του ανταγωνισμού. Αλλά καθώς ε, αυτά γίνονται από ευρωπαϊκά έργα, νομίζω πως αυτό θα μας ωφελήσει. Τέλος. Αν κατα... θα σας διαβεβαιώσω ότι στόχοι του Σικάγο να διατηρηθεί η ε, ζωντανή αμυντική βιομηχανία τους, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλιστεί η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της συμμαχικής διοίκησης μετασχηματισμού. Σας ευχαριστούμε αρχαία μου. Θα δώσω το λόγο στη συνέχεια στους συναδέλφους. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα pooling and sharing, σε μια προκλητική ερώτηση. Πολλά λέμε για τη συνένωση αυτή και εκείνη χρήση των πόρων. Αλλά τι μπορούμε να περιμένουμε από μια τέτοια προσπάθεια συνένωσης και κοινή χρήση των πόρων. Και σε ποιους τομείς κατά τη γνώμη σας αναμένουμε τις πιο γρήγορες και εντυπωσιακέ πρόοδους και τα σημαντικότερα επιτεύγματα. Ο Γιαν Πάσκου ζήτησε το λόγο. Well, thank you very much for the... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω πως όσο πλησιάζουμε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αρχίζουμε, αρχίζουν να αποκτούν ουσία τα πράγματα και νομίζω πως θα έχουμε μια ημερήσια διάταξη η οποία θα πρέπει να συζητηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν δεν θα είναι τόσο γραφειοκρατική αυτή η συνάντηση. Έχω δύο ερωτήσεις τώρα. Η πρώτη αφορά το ότι ε, καθώς ε, αποχωρούμε από το Αφγανιστάν ξέρετε πως ε, το ΝΑΤΟ θα μειώσει τη στρατιωτική του παρουσία θα έχει πολιτική παρουσία που μάλλον θα πρέπει να αυξηθεί το ίδιο αν δείτε και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείτε πως η πολιτική παρουσία ήταν ούτως ή μεγαλύτερη και η στρατιωτική παρουσία μικρότερη αλλά με βάση τα όσα συνέβησαν στην Αφρική και τα όσα μάλλον μας περιμένουν σε άλλους τομείς και σε άλλα σημεία της Αφρικής πρέπει να αυξήσουμε νομίζω λίγο τη στρατιωτική μας παρουσία. Οπότε και οι δύο οργανισμοί θα φτάσουν να έχουν την ίδια αναλογία θα έλεγα στρατιωτικής και μη παρουσίας. Και δεδομένου αυτού του σεναρίου μπορούμε να πούμε πως συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι ένα είδος pooling and sharing μεταξύ των δύο οργανισμών. Και δείτε πως θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Δεύτερο ερώτημα. Τώρα υπάρχει μια επιχειρησιακή εμπειρία. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, ε, αλλά τώρα φεύγουμε από το Αφγανιστάν και μειώνονται αυτές οι δυνατότητες. Ε, θα έχουμε όμως προκλήσεις και πρέπει να αυξηθούν οι κοινέ ασκήσεις. Αλλά με περιορισμένους προπολογισμού και, και στο μέλλον μειωμένους μπορούμε πραγματικά να θεωρήσουμε πως ε, θα αναπληρωθεί η επιχειρησιακή πείρα με τις εξετάσεις, με τις ασκήσεις, με συγχωρείτε. ή θα έχουμε λιγότερη επιχειρησιακή εμπειρία. Ευχαριστώ, Αντρίου Ευχαριστώ, καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Όλοι ξέρουμε το τι πρέπει να γίνει. Αλλά είμαι επιφυλακτικός ε, για το εάν δρομολογείται αυτό. και δεδομένου ότι θα έχουμε και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο είμαι σίγουρος πως τεχνικές προετοιμασίες για α, την συνεργασία και τις συζητήσεις για τις α, στρατιωτικές δυνατότητες προχωράει καλά αλλά δεν ξέρω εάν η φιλοδοξία που επιδεικνύουν οι πρωθυπουργοί και πρόεδροι και καγκελάροι στο σύνολό τους ε, επαρκεί. για να δημιουργήσει δηλαδή μια κοινή αίσθηση ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οπότε, κατά μία έννοια το ερώτημά μου είναι το εξής. Ε... Για ποιο λόγο αναπτύσσουμε τις ε, στρατιωτικές μας δυνατότητες. Ξέρουμε. Ειδικά στην εποχή μετά το Αφγανιστάν το ανέφερε ο κύριος Πάσκο. Μίλησε για αποχώρηση από το Αφγανιστάν. ε, ε δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως θα αποσυρθεί το ΝΑΤΟ και η Δύση από το Αφγανιστάν και θα έχουν την αίσθηση πως έκαναν καλά τη δουλειά τους και θα είναι και ικανοποιημένοι. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα αυτοπεποίθησης και στρατηγικής κατεύθυνσης και βεβαίως ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κάνει κάτι για να διορθώσει αυτή την κατάσταση αλλά καταλάβατε ήδη πως έχω τις επιφυλάξεις μου και θα ήθελα να ακούσω την άποψη των δύο διακεκριμένων ομιλητών μας και ως ε, ένα επιπρόσθετο ερώτημα θεωρείτε πως μια πρόσκληση στον Πρωθυπουργό τον κύριο Ερντογάν ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι κάτι το λογικό. Και άλλη μία ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Ε, ήρθα σε επαφή με Βρετανούς υπουργούς, όπως είναι λογικό για αυτό το ζήτημα και για άλλα, και λένε πως ε, δεν είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Ε, όπως εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να κάνουν. Εκτός αν αρχίσει να έχει πραγματικά αυτά αποτελέσματα. Και φαίνεται πως εδώ πέρα έχουμε βεβαίως ένα φαύλο κύκλο. Γιατί η υπηρεσία δεν έχει τους κατάλληλους πόρους και την κατάλληλη οικονομική στήριξη και μετά θα είναι δύσκολο βεβαίως να επιδείξει και έργο. Δεν έχω εγώ κάποια απάντηση πέραν από την αλλαγή κατεύθυνσης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, κάτι το οποίο όμως δεν το μπορούμε να το καταφέρουμε εμείς εδώ απόψε. Αλλά θα ήθελα η κυρία Αρνό να απαντήσει σε αυτά τα οποία σας περιέγραψα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κρόμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα του Πρόεδρου. Ξέρουμε πως το pooling and sharing είναι η προφανής απάντηση στο ζήτημα των πόρων και των δυνατών, δυνατοτήτων. Αλλά από την άλλη, στο ζήτημα της αυτοπεποίθησης υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά θα ήθελα εγώ να μου εξηγήσετε συγκεκριμένα το θέμα αυτό. Ξέρω πως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είχε 300 προτάσεις για το pooling and sharing και μόνο 11 από αυτές εφαρμόζονται. Οπότε το ερώτημά μου είναι, οι 290 οι υπόλοιπες, τι πρόβλημα είχαν, γιατί δεν εφαρμόστηκαν, τι επιχειρήματα ε, χρησιμοποιήθηκαν για να μην γίνουν τα υπόλοιπα έργα, για να ξέρουμε και λίγα πράγματα παραπάνω. Δεύτερο ερώτημα. Αφορά τον αντίκτυπο στις ΙΠΑ. Λένε πως οι δεν θα πληρώσουν για το 80% των νέων δυνατοτήτων. Και μια που στρέφονται προς τον ε, ειρηνικό πλέον είπα. Τι σημαίνει αυτό για την δουλειά σας, στους οργανισμούς σας. Τι άλλο αλλάζει. Πέρα από το ζήτημα, που είπαμε, της ε, πρόσκτησης ε, δυνατοτήτων. Ευχαριστώ κυρία Παναγιώτοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους δύο καλεσμένους για τις πολύ Καλέ σα παρουσιάσει. Πέρα πέρασε τη γλώσσα του Σέξπιρ, όπω είπε και ο φτέραρχο. Έχουμε όλο και πιο περίπλοκε ε, και απαιτητικέ προκλήσει ε, στην άμυνα και την ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα περικόπτουμε τι αμυντικέ δαπάνε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπου για βελτιστοποίηση των δαπανών, χωρί όμω ε, να μειώνουμε, να υποβαθμίζουμε την ασφάλεια. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα πρωτοβουλίε όπω το pooling and sharing, τη συνένωση δηλαδή και την κοινή χρήση των πόρων και την άμυνα με το Σύνοδο Κορυφή του Δεκεμβρίου που θα επικεντρωθεί και στην άμυνα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια αναθεώρηση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε έναν στρατηγικό ανασχεδιασμό και ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για μια λευκή βίβλο για την άμυνα και τις στρατιωτικές μας δυνατότητες και να επιδιώξουμε καλύτερες και περισσότερες συνέργειες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ε, ρωτώ λοιπόν τους καλεσμένους μας, ποια είναι η γνώμη σας σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα και τη χρησιμότητα μιας τέτοιας λευκής βίβλου. Πιστεύετε ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγκληση σε ό,τι αφορά μία κρεμότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που είναι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλε ερωτήσεις προς το παρόν. κυρία Αρνού και μετά εσείς στρατηγέ μου με τη σειρά που επιθυμείτε. I uh, just start with the, last question. Ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα. Τόνισα νομίζω στην εισαγωγή μου την ανάγκη και συμφωνώ πλήρως μαζί σας πως υπάρχει μία ανάγκη να υπάρξει ένα όραμα για το μέλλον εάν πραγματικά θέλουμε να έχουμε μία μακροπρόθεσμη έξυπνη άμυνα ή αυτό το pulling and sharing. Δεν ξέρω τώρα αν το καλύτερο μέσο γι' αυτό είναι μια λευκή βίβλωση ή κάτι τέτοιο, δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτό το οποίο ξέρω είναι πως για το ΝΑΤΟ υπήρξε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική η οποία είπε πως έχουμε τρεις αποστολές συλλογική άμυνα αντιμετώπιση κρίσεων και συνεργασία στην ε, ασφάλεια και μετά ε, είπαμε ποιες δυνατότητες χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε αυτές τις αποστολές. Βεβαίω, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που θα θέλαμε λόγω των μειώσεων νομίζω πως καλύτερο είναι να έχουμε κατά νου ένα όραμα ξέροντας βεβαίως πως δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον αλλά πρέπει ε, να έχουμε δυνατότητες για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και βεβαίως να αφαιρθώ σε αυτά τα οποία είπατε για τα πιο υποσχόμενα σημεία. Πρώτα απ' όλα, σημαντικό ήταν να δούμε το τι, και για μένα ήταν ενδιαφέρον, χάρη, να εφαρμόσουμε το τι έπρεπε να γίνει συγκεκριμένα στον τομέα του εναέριου ανεφοδιασμού. Και πράγματι θα βελτιωθεί. Ε, θα βελτιωθούν οι δυνατότητες ε, στην Ευρώπη και είναι μια ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές χώρες και για άλλες να συνεργαστούν προς όφελος της Ευρώπης και της ε, συμμαχίας. Και είναι νομίζω και μια σημαντική αποστολή για τη βιομηχανία. Ένας άλλος τομέας όπου ε, έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτό, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Γιατί αυτό. Γιατί μέχρι στιγμής αυτά που χρησιμοποιούμε έχουν αναπτυχθεί πριν από 10-20 χρόνια και τώρα έχουμε την ευκαιρία να εφεύρουμε μια επανδρομένα αεροσκάφη για το μέλλον που θα συμμετέχουν και σε πολιτικές αποστολές και θα εκμεταλλευτούν πλήρως την νέα τεχνολογία και επιπροσθέντως θα έχουν μια διπλή χρήση κυρίως για στρατιωτικές εφαρμογές αλλά και για πολιτικές. Και γνωρίζετε πως ε, συνεχώς αυξάνονται οι χρήσεις αυτών των μέσων για να βελτιωθεί η ασφάλεια, έλεγχος μεγάλων περιοχών, θαλασσιών και χερσαίων. Και τέλος, αυτό το οποίο μπορεί να βελτιωθεί δραματικά και έχει μεγάλη σημασία για το προσεχές μέλλον είναι η εκπαίδευση των ε, στρατευμάτων μας. Ξέρουμε πως η αποτελεσματικότητά μας σήμερα είναι αποτέλεσμα της ε, εκπαίδευσης που έχει γίνει και στην εκπαίδευση ε, υπάρχουν πολύ και διαφορετικοί τρόποι οι χώρες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να ομαδοποιήσουν την εκπαίδευση για να έχουν τις πιο αποτελεσματικές δυνατότητες και αυτό πρέπει να γίνει και με μια πιο ευρωπαϊκή ε, προοπτική ή με μια πιο υπερατλαντική λογική. Αυτή θα έλεγα πως είναι η πιο πολλά υποσχόμενη τομής ε, μέσω πρόθεσμα. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω πρώτα στην τελευταία ερώτηση γιατί πιθανότατα είμαι στη μειοψηφία και μιλώ περισσότερο σε προσωπική βάση, γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει γνώμη του οργανισμού αμήνης όσον αφορά κάτι τέτοιο. Ιδανικά και πνευματικά θα ήταν πολύ καλό να έχουμε ένα κοινό λευκό βιβλίο. Και εγώ δεν είμαι θεωρητικός καταρχήν. Τα πρώτα χρόνια μάλλον τις πρώτες δεκαετίες της ζωής μου γράφοντας διάφορα έγγραφα και το ευχαριστιόμουν και γι' αυτό και δεν είμαι πολύ επιφυλακτική. Το να φτιάξουμε τώρα μια τέτοια, να κάνουμε τώρα ένα εγχείρημα θα μπορούσε να μας διαιρέσει, να είναι πολύ καδημαϊκό. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε, δεν χρειάζεται να ορίσουμε κάποιο μέσο να ορίσουμε μια απειλή ας πούμε, συγκεκριμένη που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε 30 χρόνια. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε κατά τη γνώμη μου είναι να ε, στιάσουμε την προσοχή όχι σε έναν ορισμό του τι θα πρέπει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα πρέπει να κάνουμε στο ΝΑΤΟ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να αρπάξουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν τις δυνατότητες, τις ικανότητες τις δυτικές για οποιοδήποτε είδους δράση για, και, ενώ και στρατιωτική δράση που θα μπορούν να θέλουν να κάνουν επιχείρηση. Είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε πλαίσιο ΝΑΤΟ, είτε σε πλαίσιο Ένωσης. Δεν προβλέπω για αύριο μεθαύριο μια άσκηση όπου τα κράτη-μέλη μας θα είναι επιτυχή είτε θέλουν να κάνουν εθνική εθνικά στρατιωτικά ή στο ΝΑΤΟ ή στην Ένωση. Κάτι τέτοιο λοιπόν όπως, θα, είπα θα, είναι, ε, θα μας διχάσει και θα είναι επίσης ένα άλοθη για να μην δουλέψουμε πάνω στο συντονισμό των ικανοτήτων μας. Και όπως είπε και ο Πτέραρχος, ε, υπάρχει μια στρατηγική τέτοια έννοια στο ΝΑΤΟ και δεν θα είναι και τόσο διαφορετικές οι ικανότητες που θέλουμε να αναπτύξουμε, ώστε να ξέρουμε χοντρικά πού κατευθυνόμαστε όσον αφορά τις αρνητικές ικανότητες. Επίσης, αυτό που θα ήταν χρήσιμο είναι τα κάτι μέλη να φτιάξουν ένα έχουν ήδη ένα λευκό βιβλίο και θα έπρεπε να έχουμε ε, συντονισμό και συνεννόηση συγγράφοντα κάτι τέτοιο. Είχα το προνόμιο να συμμετέχω στη Γαλλική Αντίστοιχη Επιτροπή για το ε, ε, Λευκό Βιβλίο και ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μήνης για να υπάρξει ένα συντονισμό, να, δούμε, να δώσουμε συμβουλές, εμπειρογνωμοσύνη, να τους πούμε τι κάνουν οι άλλοι, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το μέσο που έχουν ώστε να υπάρχει καλύτερη ο συντονισμός για το λευκό βιβλίο και, στα συμπερα... για τα συμπεράσματα του λευκού ε, βιβλίου. Να πούμε, ας πούμε, τώρα αποφασίσαμε αυτό ή μάλλον πριν αποφασίσω αυτό, τι είδους ικανότητες μπορώ να έχω από κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ή αν έχω τις τάδε ικανότητες σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν πια αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είμαι υπέρ αυτής της άσκησης που μας δόθηκε ως μια αξιολόγηση επί τη βάση του κώδικα διοντολογίας για το πού βρίσκονται τα διάφορα κράτη-μέλη και είμαι υπέρ αυτής, αυτής της επαφής ως ένα πρώτο βήμα για την επεξεργασία του Λευκού Βιβλίου από τα κράτη-μέλη και φυσικά η EDA είναι έτοιμη να το στηρίξει αυτό. ώστε έτσι στη συνέχεια να είμαστε λιγότεροι, λιγότερο επιφυλακτικοί για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού βιβλίου. Αλλά μετά από αυτό το πρώτο βήμα συνεννόησης επαφών και λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα γίνονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Για να επανέλθω στο ερώτημα 1 του Προέδρου για την συγκέντρωση και κοινή χρήση, ποια είναι τα αποτελέσματα. Υπάρχουν προφανή αποτελέσματα σε ορισμένους τομείς που είναι νομίζω στρατηγική σημασία. Αν δούμε τις ε, τηλεπικοινωνίες, δορυφορικέ τηλεπικοινωνίες, έχουμε φτιάξει μια μονάδα στην, στον οργανισμό μας για την ε, για την κοινή χρήση και διάθεση σε όλα τα κράτη-μέλη των συμβάσεων που έχουμε. Δηλαδή έτσι έχουμε καλύτερες τιμές, καλύτερες ε, όρους διαθεσιμότητας για τις ώρες επικοινωνίας μέσω δορυφόρου. Και ξέρουμε βέβαια και πάντοτε υπό την αίρεση των, της του Στατηγού ότι οι επικοινωνίες μέσω δορυφόρου είναι θέμα κλειδί. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τόσο μεγαλύτερη συγκέντρωση πληροφοριών έχουμε και άρα τόσο πιο σημαντική είναι και η μετάδοση των δεδομένων μέσω δορυφόρου. Και γι' αυτό και κάναμε αυτήν την ε, συγκέντρωση της σύμβασης. Το ανάλυσαν και οι Υπουργοί το, και το ΕΝΕ, αλλά πρέπει να δουλέψουμε για την μελλοντική γενεά δορυφόρων ε, τηλεπικοινωνιών. Δεύτερο παράδειγμα είναι η θαλάσσια εποπτεία που έχουμε πάλι κοινή χρήση του χώρου θαλάσσιας εποπτείας ανάμεσα στα 15 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε με δυνατότητα ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών και άρα αντιμετώπισης διαφόρων περιστάσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις του ναυτικού στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν άλλοι τομείς που ήδη αναφέραμε και που ο κτέραρχος τους ανέφερε στον τομέα ας πούμε Ε, των ασκήσεων για τα πληρώματα ελικοπτέρων. Αυτό μας επέτρεψε να αναπτύξουμε πληρώματα πολύ καλά εκπαιδευμένα στο Αφγανιστάν. Τα κάτι μέλη που ήθελαν να στείλουν ελικόπτερα στο Αφγανιστάν είχαν εκπαιδευμένα πληρώματα. Έπειτα είχαμε συγκέντρωση και κοινή χρήση με τον ΝΑΤΟ, ε, άρα ένα τμήμα που πάει στον κύριο Πάσκου και έπειτα βελτιώθηκε και η ασφάλεια των πληρωμάτων. Και πέρα από τα ελικόπτερα είναι κάτι που θα κάνουμε από εδώ και μπρος και για τα αεροπλάνα και για μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων. Και ελπίζω το επόμενο παράδειγμα που θα μπορέσω να σας αναφέρω μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι ο αναέριος για τον κύριο Πάσκο για το συγκέντρωση και κοινή χρήση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς ήδη το ανέφερα ότι κατά τη γνώμη μου αυτή η δυνατότητα να μπορούμε να δουλέψουμε στο ΝΑΤΟ την πτυχή του στρατικού εξοπλισμού και, εδώ, και, στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό το πλήρωμα είναι ένα είδος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε pooling and sharing, πάντως είναι μοιρασιά των ε, καθηκόντων. Το ίδιο και όταν μπορούμε να δουλέψουμε ε, ας πούμε σε ένα σεμινάριο στον οργανισμό μας ε, για την καταπολέμηση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και το, τα όσα κάνουμε εμείς τα χρησιμοποιεί και η ISAF έχουμε πραγματική κοινή χρήση ανάμεσα στην Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον ε, ιατρικό εξοπλισμό. Πάντως, Αυτό που κάνουμε είναι ότι επιλέγουμε ένα πλαίσιο για να κάνουμε μια δράση, αλλά οι ικανότητες που απορρέουν από αυτό είναι απολύτως στη διάθεση του ΝΑΤΟ, αλλά και στη διάθεση των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο και το ίδιο ασχεί και αντιστρόφως ανάλογα στο πλαίσιο της Smart Defense, της εφιούς άμυνας. Για την πολύ δύσκολη ερώτηση του κυρίου Νταφ. Για, για το κατά πόσο θα φανούν στο ύψος των περιστάσεων ε, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής ως προς τις προσδοκίες που έχουμε δεν έχουμε το αυριανό σενάριο. Ετοιμάζουμε τις δυνατότητές μας ε, για την επόμενη 20 ετία, 30 ετία. Δεν υπάρχει αξιόπιστο σενάριο που δεν θα περιλαμβάνει και στρατιωτικό σκέλος. Θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα και στρατιωτικής ε, άσκησης ε, εξουσίας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν και για τις αυριανές μας δυνατότητες με υψηλότερο βαθμό τεχνολογίας για να είμαστε και πιο, ευπροσάρμοστοι. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις μελλοντικές απειλές και τους αυριανούς μας εχθρούς, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και απειλές και κατά πάσα πιθανότητα και εχθροί. Οπότε από τώρα θα πρέπει να ετοιμάσουμε τις δυνατότητές μας με το υψηλότερο επίπεδο της αυριανής προηγμένης τεχνολογίας. Και νομίζω ότι γνωρίζουμε προς τα που θα πρέπει να στραφούμε ως προς τις τεχνολογίες και τις δυνατότητές μας. Προς το παρόν πάντως γνωρίζουμε και τις αδυναμίες μας. Και δεν θα είναι και πολύ διαφορετικές από τις μελλοντικέ, γιατί οι σημερινές μας αδυναμίες είναι ίδιες με τις αδυναμίες που είχαμε πριν από μία δεκαετία, πριν δηλαδή τις επιχειρήσεις ε, στην πρώην Οικοσλαβία. σε ό,τι αφορά την ε, πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου θα το αφήνω στον Πρόεδρο. Στον Πρόεδρο της Υποεπιτροπής. Σας ό,τι αφορά τις, ε, τους πόρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, την ερώτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να, είμαι και πιο, να είμαι ο οργανισμός μας και πιο αποτελεσματικός αν ε, δεν αναλωνόμασταν ε, σε αυτόν τον αγώνα να αναπτύξουμε αυτούς τους ε, ισχνούς πόρους που έχουμε. Πάντως έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο υπουργών και χρειαζόμαστε ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων. Πιστεύω πάντως ότι υπάρχει το θέμα του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, αλλά πιστεύω ακράδαντα ε, δεδομένη της ε, δημοσιονομική κατάστασης των κρατών μελών που είναι και παράμετρος των δράσεών μας, το γεγονό ότι έχουμε πια την πραγματικότητα του pooling and sharing. Δεν έχουμε μια, πια μόνο την εμπειρογνωμοσύνη του ΕΝΤΑ, αλλά τη δυνατότητα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και τα έργα θα τα κάνουν τα κράτη-μέλη. Εμείς με τους πόρους μας θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποια προγράμματα στα κράτη-μέλη, όπως τον ενέργειο εφοδιασμό σε καύσιμα, αλλά η απόφαση για τις αγορές, για τις προμήθειες, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ένα 2% επιπλέον που θα αλλάξει την απόφαση. Πάντως για, μας ο βασικός, για μένα ο βασικός παράγοντας είναι τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να επενδύσουν στις δράσεις, στις αγορές, στην κατάρτιση με βάση τις δικές μας προτάσεις. Δεν λέω ότι το θέμα του προπολογισμού δεν είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε πρώτα συγκεκριμένο προπολογισμό για συγκεκριμένες δράσεις που αποφάσισαν να αναλάβουν τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι πρακτικές αποφάσεις των κρατών μελών, ώστε να εφαρμόζουν οι προτάσεις του ΕΝΤΑ και τα κράτη-μέλη να επενδύουν ώστε να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας όπως τον αέριο εφοδιασμό σε καύσιμα. <laughs> Τώρα, τι, ποια είναι τα κενά, ποιες είναι οι αδυναμίες ε, στο pooling and sharing, τη συνένωση και την κοινή χρήση των πόρων. Εγώ όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ανέλαβα την πρωτοβουλία και πήρα την προ... και υπέβαλα την πρόταση να προτείνω στα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν σε λίγες προτεραιότητες. Και αυτά που προτείνουμε είναι οι προτάσεις μας για άμεση δράση, με βάση την οξύτητα και τη σοβαρότητα των προβλημάτων και με βάση το κατά πόσο είναι εφικτές οι προτάσεις. Το πρώτο θέμα φυσικά είναι η εμπιστοσύνη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μέλων. Η συνεργασία προϋποθέτει τέτοια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και αυτό λαμβάνεται υπόψη στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος και από τη που θέλουν τα κράτη-μέλη μια δυνατότητα να μπορούν να τη χρειάζονται να την επικαλεστούν. Ε, μερικά κράτη-μέλη ε, αυτό σημαίνει αυτόματη απόκριση των εταίρων και για ορισμένα σημαίνει απλώς ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα του σεβασμού των πολιτικών και των κοινοβουλευτικών αποφάσεων. Τώρα, όταν μιλούμε για, για σχέδια, προγράμματα pooling and sharing και για ανάπτυξη των δυνατοτήτων, μιλήσαμε για τις εναέριες μεταφορές, την εναέρια, τον εναέριο ενεφοδιασμό και έχουμε κάποιες αποφάσεις που ενεκρίθηκαν από τη EATC και μπορούμε να πούμε στα κράτη-μέλη ότι υπάρχει μια λύση. Μπορείτε να έχετε αμοιβή εμπιστοσύνη και ότι θα έχετε στη διάθεση σε αυτές τις δυνατότητες όταν τις χρειάζεστε. Ένα άλλο εμπόδιο είναι ότι για πολλές δυνατότητες τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επενδύσουν. Και είναι δύσκολη καιρή για επενδύσεις, είτε εξαιτία των περικοπών των δαπανών, είτε γιατί τα κράτη-μέλη είναι σε φάση που είναι δέκτες δυνατοτήτων που είχαν σχεδιάσει το παρελθόν. Εξαρτάται σε ποιο κύκλο βρίσκονται δηλαδή, αν είναι δέκτες ή πάροχοι των δυνατοτήτων. Και αυτή που είναι στη φάση του δέκτη είναι δύσκολο να ξεκινήσουν νέα προγράμματα. Και από αυτό αυτή την άποψη θα πρέπει να δούμε αν είναι ρεαλιστικό αυτό το παράθυρο της ευκαιρίας. Επίσης θα πρέπει να πείσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα που θα πρέπει να δείξουν ότι ήταν επιτυχή. Μόνο με επιτυχίες θα πείσουμε τους άλλους. Δεν είναι εύκολο να πείσουμε τους υπουργούς σε πολιτικό επίπεδο, αλλά τα έμπρακτα αποτελέσματα και η επιτυχία σε πρακτικό επίπεδο θα είναι η καλύτερη απόδειξη. Και έτσι θα πείσουμε όχι μόνο τα ανώτατα του υπουργού, αλλά και όλο το μηχανισμό των Υπουργείων Άμυνα. Γιατί τα Υπουργεία Άμυνας, άμυνας μέχρι στιγμής δεν ε, φτιάχτηκαν για συνεργασία. Η συνεργασία είναι κάτι που θα κατακτηθεί σταδιακά και με βάση την εμπιστοσύνη που θα δημιουργηθεί από τις κοινέ επιτυχίες. Προσπάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Επανέλθω σε δύο κρίσιμα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ. Θέλω να ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα. Για το Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ δεν αποσύρεται από το Αφγανιστάν η αποστολή θα αλλάξει και θα συζητηθεί αύριο και μεθαύριο επί τη ευκαιρία από τους υπουργούς οι οποίοι λογικά θα συμφωνήσουν σε ένα νέο επιχειρησιακό πλαίσιο για την αποστολή η οποία θα είναι εκπαιδευτική και επικουρική των Αφγανικών δυνάμεων και σε επίπεδο συμβούλων. Θα υπάρχει όμως ένα ικανό στοιχείο, μια μελλοντική αποστολή στο Αφγανιστάν και προφανώς υπάρχει θέληση για μια πιο ε, συνολική προσέγγιση και περισσότερη συνεργασία. Παρ' όλα αυτά με το Αφγανιστάν ε, λογικό είναι θα μειωθεί ε, το εύρος των επιχειρήσεων. δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά παρόλα αυτά αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Και μην ξεχνάμε πως ε, μετασχηματισμός των δυνάμεων είναι πολλά υποσχόμενος. Η διαλειτουργικότητα των δυνάμεων και μέσω τεχνολογικών μέτρων και μέσω κοινή εκπαίδευση ε, και βελτίωσης εκπαίδευση ε, και ασκήσεων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και πραγματικά προσπαθούμε για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που έχουμε είτε υπό την, ευκαιρία, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ είτε με κάποιο άλλο σχήμα. Και υπάρχει επίσης και μια πτυχή τεχνολογική και βιομηχανική. Οπότε είναι κάτι το οποίο ε, για το μέλλον έχει ε, σοβαρές προοπτικές και δεν αφορά τον Άτομο μόνο, σημαίνει η σύνδεση των δυνάμεων με τις χώρες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΝΑΤΟ, με όσο δυνατόν περισσότερους. Αυτά από εμένα. Για τον άξονα τον είπα προς την Ασία. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά βέβαια, αλλά θα έλεγα πως από τη σκοπιά τον είπα. Μια που ζω και εργάζομαι εκεί, μπορώ να σου πω πως υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες των Αμερικανών συμμάχων μας, ε, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να γίνουν περισσότερο πάροχοι και όχι καταναλωτές ασφαλείας και τεράστιες προσδοκίες οι ευρωπαϊκές χώρες να επιδείξουν την θέλησή τους για να αυξήσουν τις δικές τους δυνατότητες σε πλήρη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, αλλά πάντα με τη βούληση να έχουμε θα έλεγα συγκεκριμένη συμμετοχή στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ξεκάθαρο στη ΣΥΠΑ. Κάθε εβδομάδα έχω επαφές στην Ουάσιγκτον με κάποιους που μου λένε πρέπει επιτέλους οι ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν κάτι ε, και υπάρχει θα έλεγα ένα παράθυρο ευκαιρίας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους ε, μπορεί να αποστείλει ένα μήνυμα προς τις ΕΠΑ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πτεραρχή. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω θερμά τους συναδέλφους από την Ολλανδική Βουλή που μας έκανα την τιμή να έρθουν στην Υποεπιτροπή ε, της ε, άμυνας, ε, ασφάλειας και άμυνας από την, Ολλανδική, από την Επιτροπή Άμυνας της Ολλανδικής Βουλής. Γνωρίζετε την κυρία Αρνού, την Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και τον πτέραρχο Παλομέρος που είναι ανώτατος διοικητής της Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού. Συζητούμε τα θέματα άμυνας εν ώψη του Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου. Θα δώσω το λόγο στον Άντριου Νταφ, Μία σύντομη ερώτηση για τη Λευκή Βίβλο. Η κυρία Αρνού μας είπε ότι θα ήταν χρήσιμη μία αλληλεπίδραση και σχετισμό με τις εθνικές ε, στρατηγικές και της αναθεώρησης της άμυνας. Πιστεύετε ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να προωθηθεί με τη δημιουργία ε, ενός κοινού προτύπου για τις ε, στρατηγικές αναθεώρησεις ώστε όλοι οι Υπουργοί Άμυνας με τον ίδιο τρόπο με βάση κοινό, κοινή μεθοδολογία να προβαίνουν στην αναθεώρηση και να κάνουν την αξιολόγηση. Μάλιστα, κάτι τέτοιο θα μπορούσαν να το κάνουν και ταυτόχρονα, γιατί όχι. Euh, Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, κύριε Αρνού, αναφερθήκατε στην ομιλία σας και στο θέμα αυτό. Τι ευέλεια θα πρέπει να έχει μια προσπάθεια υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Και με ποιο τρόπο θα μπορούσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας να διευκολύνει τις επενδύσεις αυτών των επιχειρήσεων ή μάλλον προς επιχειρήσεις αυτές. Τι μεθοδολογία μπορούν να ακολουθούν οι επιχειρήσεις, να στρέφονται απευθείας σε εσά, να περνούν από τα κράτη-μέλη, πολύ καινοτόμα ιδέα και πολλά υποσχόμενη. Και μια πιο πολιτική υφής ερώτηση. Και για το Smart Defense και για το Pooling and Sharing, πώς πιστεύετε σε μια τέτοια χαλεπή περίοδο μπορούμε να αποτρέψουμε την αποσύνδεση κάποιων μικρών χωρών, κυρίως ό,τι αφορά την επιθυμία επενδύσεων στην άμυνα, να μην τις χάσουμε στην πορεία. Και παρά το Smart Defense και παρά το Pooling and Sharing, μήπως έχουμε μια ειδίκευση, εξειδίκευση των προσπαθειών της άμυνας με ορισμένες μονοχώρες που θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια ενώ άλλες θα μένουν στην πορεία πίσω. Δηλαδή δεν θα ενδιαφέρονται στο μέλλον για συμμετοχή ούτε καν σε κοινά προγράμματα. Πιστεύετε ότι είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος είναι μόνο δεν πρόκειται να κατονομάσω συγκεκριμένες χώρες, αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να απειλήσει την ομοιογένεια και την ομοιομορφία και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα στρατιωτικά και άμυνας. Uh, να ξεκινήσουμε ίσως με την ε, ιδέα του κυρίου Νταφ. Νομίζω ότι να έχουμε πιο κοινά χρονοδιαγράμματα θα ήταν πολύ χρήσιμο. Έχουμε ένα κρατος μέλος που φτιάχνει το Λευκό Βιβλίο, ένα άλλο που φτιάχνει την αναθεώρηση κτλ. Πάντως, αν υπήρχε μεγαλύτερη σύγκληση στα χρονοδιαγράμματα, αν και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, ξέρουμε ότι συνδέεται με τα πολιτικά χρονοδιαγράμματα, ωστόσο, όπως και τα παιδιτικά φόρουμ. Πάντως, όσο πιο κοντά ε, μπορούσαν να είναι τα χρονοδιαγράμματα, τόσο το καλύτερο τώρα. Κοινέ ε, ιδέε, ναι, θα ήταν ιδανικό για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Ταυτόχρονα βλέπουμε μέσω των συγκεκριμένων άσκησης στις οποίες συμμετείχα, βεβαίως τα δόγματα της δικής σας του δικού σας λευκού βιβλίου ε, σχετίζεται με τις αποστολές του στρατού σας και θα ήταν πολύ διαφορετικό από το ένα κράτος στο άλλο. Αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινά στοιχεία και ίσως κάποια ευελιξία, γιατί για κάποια κράτη ας πούμε υπάρχει μεγαλύτερος ρόλο για το ναυτικό ή για την αεροπορία, περισσότερος χώρος για πολιτική υπηρεσία. Με περιπτώσει θα υπήρχαν διάφορα ε, σημεία, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε σε ευελιξία πιο συγκεκριμένα για τα κράτη-μέλη. Και κάτι ακόμα που ξέχασα γιατί ο Πτέρος Παλωμερός το ανέφερε πριν τη σημασία τη σύνδεση με τη ΣΥΠΑ. Ο αντίκτυπος του οργανισμού είναι πολύ απλός, πολύ μεγάλη στήριξη για οτιδήποτε κάνουμε. Είμαστε πολύ μεγάλος οργανισμός και μόνο να φανταστεί κανείς τον προπολογισμό που έχουμε σε σύγκριση με τα αμερικανικά στάνταρ, αυτό τους ενδιαφέρει και το να το στηρίξουν Είχαμε προσκλήσει από τα κρατημέλη, από τα έθνη για να συμμετέχουν στις ασκήσεις, πολυεθνικές ασκήσεις σχεδια, αμυντικού σχεδιασμού ε, και για τον εναέριο ανεφοδιασμό. Ήθελαν να επιτύχουμε και θα ήταν και πολύ αυστηρή αν αποτύχουμε. Εξέφρασαν τη στήριξή τους στο ΣΥΚΑΟ και αναμένουν τα αποτελέσματα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στηρίζουν ε, λοιπόν αυτές τις προσδοκίες. Τώρα αν δεν υλοποιηθούν δεν θα είναι καλό για μας αυτό. Και μάλιστα όπως είπε και το ίδιο το Πεντάγωνο θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο έπειτα εκείνους να έχουν τον προϋπολογισμό για την διατλαντική αλληλική αν δεν δείξουμε κανένα σημάδι βούλησης και αποτελέσματος. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι πως πρόκειται για πολύ σημαντικό τμήμα του τεχνολογικού και βιομηχανικού μας κεφαλαίου. Επίσης αυτό οδηγεί στο ότι όλα τα κράτη-μέλη αισθάνονται απόλυτα δεσμευμένα στα όσα μπορούμε να κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Προτείναμε στα κράτη-μέλη μα ένα σχέδιο δράση στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μάλιστα εμπνευστήκαμε πολύ από το τι κάνουν σε εθνικό επίπεδο για να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ολόκληρη σειρά δράσεων λοιπόν προτείνεται και που φυσικά σε πολλέ περιπτώσει είναι περισσότερο παροτρύνσει. Δεν πρόκειται για κάτι το ρυθμιστικό, πρόκειται για διευκολύνσεις ώστε οι μικρομεσαίες να μπορέσουν να ωφεληθούν από τα αμυντικά προγράμματα και από τι διάφορε δραστηριότητε. Επί τη βάση των συζητήσεών μα με του συναδέλφου ε, τη Κομισιόν που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ε, μικρομεσαίων, ε, είμαι πεπισμένη ότι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί αν εστιάσουμε την προσοχή σε συγκεκριμένε δραστηριότητε και γι' αυτό το λόγο και προτείναμε τα μη μικρά μη επανδρομένα σκάφη και την κυβερνοάμυνα γιατί είναι ένας όπου οι μικρομεσαίες μπορούν να παίξουν στη ρόλο αριστείας και να φέρουν με πολύ προστιθέμενη αξία. Όχι μόνο λοιπόν οριζόντια δράση, αλλά να το αποδείξουμε σε ε, τομείς κλειδιά όπως τα μικρά μη επανδρομένα αεροσκάφη και η κυβερνοπροστασία. Διαδικασία. Τώρα κανονικά έχουμε σχέσεις με συνδέσμους ενώσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η σύνδεση βιομηχάνων τα ρυθμίζουν όπω ε, κρίνουν. Πάντως εμείς ως Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνη θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερε επαφές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε, ερχόμαστε σε επαφή με τι Εθνικές ενώσει Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Βλέπουμε όλους τις συνδέσμους που συνδέουν διάφορα κρατημέλη. Αν θέλετε, εμεί χρησιμοποιούμε κάθε δυνατή λαβή για να έχουμε επαφέ με τι μικρομεσαίες γιατί είναι εκθέσεις στο Βερολίνο, το Λονδίνο ή το Παρίσι. Ε, βρισκόμαστε επίσης ε, στις εκθέσεις στις διάφορες εκθέσεις για να έχουμε επαφές τακτικές. Πιο συγκεκριμένα για τα διευθυντικά ταμεία Ερευνήσαμε ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη μας και τους διάφορους φορείς του, της αμήνης για να ωφεληθούν από τα ε, διευθυντικά ταμεία. Κάναμε μια μελέτη για να εντοπίσουμε ποια είναι τα κριτήρια, ποιε είναι οι διαδικασίε. Διοργανώσαμε και ατελεία με του διάφορου φορεί και θα πάμε στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν, ώστε ακόμη μια φορά να βοηθήσουμε του διάφορου φορεί και πιο συγκεκριμένα για να βρούμε χώρα στις μικρο... για τι μικρομεσαίε, για τη χρήση των διορθωτικών ταμείων και χρησιμο... συζητούμε και με την Κομισιόν για πιστώσει όπω το COSME, που είναι συγκεκριμένε γραμμέ για τι μικρομεσαίε. Και η Κομισιόν έχει δίκιο, έχει υπάρχει πρέσβης για, το, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, προχωρά χέρι με χέρι με τη Γενική Διεύθυνση για τι επιχειρήσει για να φτιάξει μέσα από ένα δίκτυο που καλύπτει όλε τι μικρομεσαίες, να ενημερώσει έτσι όσο γίνεται περισσότερο και να απαντήσει στα ερωτήματα των μικρομεσαίων στον τομέα τη Άμυνα Εν γέννη δεν τους αρέσει να λέμε άμυνα, να τους αρέσει καλύτερα να λέμε άμυνα και ασφάλεια ασφάλεια και άμυνα για την αλήθεια ότι οι δραστηριότητε του είναι ευρύτερε. Για τις μικρές χώρες και το εναπόλυα ενδιαφέροντος θα σας πω ότι γενικό αίσθημα είναι πως οι μικρές χώρες, τουλάχιστον όσο τη δράση, τη δραστηριότητα, ε, είναι απόλυτα μέσα στην διαδικασία και το λέω με μεγάλη υπεποίθηση όσον αφορά τις ε, ικανότητες. Στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνης ε, οι χώρες που ηγούνται για διάφορες δραστηριότητες είναι μικρές χώρες γιατί δεν χρειάζεται να τις πείσει κανείς για τη συνεργασία για εκείνες είναι ήδη μια εμπειρία που γνωρίζουν, ξέρουν πόσο ζωτική σημασία είναι και βρίσκω ότι όσον αφορά την συμμετοχή του στις δραστηριότητες, η συμμετοχή των μικρών χωρών είναι πολύ καλή, σε πολύ καλό επίπεδο Υπάρχει βέβαια περιθώριο βελτίωση όσον αφορά τη συμμετοχή των μεγάλων χωρών. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη πω και εδώ υπάρχει ένα ε, ρόλο καταλήτη των μεγάλων χωρών που οφείλουν να τον παίξουν και πρέπει να βελτιωθεί. Τώρα, το θέμα του προπολογισμού. Με ρωτήσατε και γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιε μικρέ χώρε που αυξάνουν τον προπολογισμό του. Φυσικά ξεκινούν από μικρά ποσά, αλλά πρέπει να δούμε την εξέλιξη. Και νομίζω πως υπάρχουν θετικά στοιχεία εξέλιξης από πλευράς ορισμένων μικρών χωρών. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να τις βοηθήσουμε, να τους δείξουμε και ότι θα έχουν ωφέλη όσον αφορά την ασφάλεια. Και άρα να λάβουμε υπόψη όλες τις επιταγές ασφαλείας τους όχι μόνο αυτές των μεγαλύτερων χωρών, βέβαια θα πρέπει να βλέπουν και κάποιο όφελος βιομηχανικό, οικονομικό και τεχνολογικό. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες. Και επίσης πρέπει να έχουν και ωφέλη όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Οι μικρές και μεσαίες χώρες λένε περισσότερο ότι χρειάζονται πραγματικές πολιτικές ασφάλειας και άμυνας, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται να δείξουμε πως υπάρχει λόγος να υπάρχουν κοινέ στρατιωτικέ ικανότητες όταν είμαστε σε ένα καθεστώς ακόμα και ουδετερότητας και μόνο η δραστηριότητα, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας μπορούν να δώσουν νομιμότητα σε έναν προϋπολογισμό αμήνης, γιατί διαφορετικά δεν είναι νομιμοποιημένος ένας τέτοιος προϋπολογισμός ιδιαίτερα στις πολιτικές ε, ουδετερότητας το γεγονός ότι υπάρχει μια ζωντανή και λειτουργούσα κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνες, είναι ένα βασικό στοιχείο ώστε οι μικρές χώρες να μπορούν να αποδείξουν την θεμητότητα, την νομιμότητα ενός ε, αμυντικού προπολογισμού. Επ' αυτού θα ήθελα να το μίσω, χωρίς να διαφωνώ, πως ε, σε πολλές χώρες που επισκεφτούμε, οι στόχοι του ΝΑΤΟ είναι οι πιο σημαντικοί από πλευρά ε, αμυντικού προπολογισμού. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή το σημείο αναφορά είναι οι δεσμεύσει ε, του ΝΑΤΟ. Όπω αυτό γίνεται μέσω τη ε, διαδικασία σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει και υπάρχει κάποιος συντονισμό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία, οπότε υπάρχει κάποιο τρόπο. για ένα κοινό όραμα και τα έργα βεβαίως έχουν κάποιες κοινέ ε, συζητήσεις, πολυμερείς συζητήσεις και μετά καταλήγουμε σε μια ισορροπία τι είναι εφικτό, ποια χώρα μπορεί να αναλάβει το κάθε καθήκον και υπάρχει μια δικασία αλλά σε τελική ανάλυση νομίζω πως ε, υπάρχουν αυτά τα πράγματα και επί τη ευκαιρία θα παρουσιαστούν και αύριο στους Υπουργούς Άμυνας. Για τις μικρότερες χώρες. Έχουμε πολλά παραδείγματα συνεργασίας. Αυτό το οποίο γνωρίζω καλύτερα είναι η ε, άμυνα, η αεροπορική των χωρών της Βαλτικής που την εξασφαλίζουν οι χώρες του ΝΑΤΟ εκ περιτροπής και έτσι δεν επενδύουν σε δικά τους μαχητικά αεροπλάνα οι χώρες αυτές. Παρόλα αυτά έχουν δικές τους δυνατότητες ε, ελέγχου και έτσι ελέγχουν τον εναέριο χώρο τους ε, χρησιμοποιώντας ε, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Είναι λοιπόν μία έξυπνη άμυνα θα έλεγα και όταν επισκέφτηκα αυτές τις χώρες είδα πως υπάρχει όρεξη για περισσότερα τέτοια αρκεί να μπορέσουμε να ορίσουμε ε, κοινά συμφέροντα και αυτό είναι το βασικό εάν οι χώρες αυτές έχουν κίνητρα γιατί θεωρούν πως είναι προς το συμφέρον τους να συνεργαστούν θα το κάνουν δεν είναι εύκολο, χρειάζεται χρόνος χρειάζεται ε, υπομονή και υπάρχουν πολλά ζητήματα και νομικά και δεν είναι τα πιο εύκολα αλλά είναι εφικτό θα έλεγα και αντιλαμβάνονται πως είναι καλύτερο να ε, σχεδιάζουν αντί να χάνουν δυνατότητες και οι μεγάλες χώρες χάνουν κάποιες δυνατότητες γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Οπότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν την νέα αυτή προσέγγιση και βεβαίω μπορεί να υπάρξει μια νέα ένας νέος σχηματισμός αλλά ε, μπορεί και οι χώρες να αναπτύξουν άλλες ε, να αναπτύξουν άλλους συνδέσμους. Θεωρώ λοιπόν πως θα έχουν ε, θα έχουμε περισσότερες τέτοιες ε, κινήσεις ε, στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Βαντάλη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Θα ήθελα να πω ότι αν θέλουμε συνένωση και κοινή χρήση θα πρέπει να έχουμε κάτι να συνενώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε από κοινού. Γιατί όλοι κάνουν περικοπές και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε λοιπόν συνένωση και κοινή χρήση, θα πρέπει πρώτα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσουμε πού θέλουμε να επενδύσουμε σε hard power ή σε soft power. Αυτό είναι θέμα απόφασης και πώς θα κάνουμε την κατανομή των καθηκόντων. Νομίζω ότι έτσι θα αποφύγουμε τα προβλήματα. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι ευθύνες έχει ο καθένας. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά ίσως πρέπει να έχουμε στρατηγική και hard power και σκληρή δύναμη και ήπιας δύναμη, soft power, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Κύριε κυρία Αρνού. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι φροντίστε να αναλάβετε επιχειρήσεις σαν αυτή και μόνοι σας. Αυτό είναι θέμα hard power. Και πρέπει να το αναλάβουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να βρούμε τα, κράτη-μέλη που θα αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες που είναι πιο μεγαλεπίβολες και αν θέλουν κάποιες μεγάλες χώρες μέλη να αντικαταστήσουν τις Ηνωμένε Πολιτείες στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να παίξουν ένα πιο καταλητικό ρόλο για να αντικαταστήσουν αυτό το 80% που μέχρι τώρα συνεισέφερε στο ΝΑΤΟ οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε και hard power και σκληρή δύναμη, όχι μόνο ήπια δύναμη. Και πιστεύω ότι και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ είναι το ίδιο, ότι soft power, ε, η ήπια δύναμη μόνη της ε, είναι ουσιαστικά δυναμία θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε και τέτοια σκληρή δύναμη. Και η πρόταση, μου λέει ο Πτέραρχος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως η καταλληλότερη οργάνωση ε, για να βρει το σωστό μείγμα μεταξύ σκληρής και ήπιας δύναμης, hard και soft power. Και εγώ πιστεύω ότι και τα δύο είδη δυνάμεις χρειάζονται στην εποχή που ζούμε. Και κατά τη γνώμη μου αυτό θα πρέπει να κάνουμε στο μέρο να βρούμε το σωστό μείγμα αυτών των δύο δυνάμεων και την ισορροπία μεταξύ τους. Γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο μορφών δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι είναι σαφή τα όρια μεταξύ του hard power και soft power σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για παράδειγμα, που αφορά κυρίω εικονικά περιστατικά. Οπότε και είναι ακόμη πιο δύσκολη η διάκριση μεταξύ των δύο. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε το πρώτο τμήμα της συνεδρίας. σα. ευχαριστούμε κύριε Πτέραρχη για την πρώτη σα παρουσία εδώ. Ε, πρώτη λέω γιατί είμαι σίγουρο ότι υπάρχει συνέχεια στις επαφέ μα και οι, οι πόρτες μας θα είναι διάπλατα ανοιχτές και είστε ευπρόσδεκτο. Το ίδιο ευπρόσδεκτη θα είναι πάντα και η κυρία Αρνού. Και Νομίζω ότι οι αρχές του 2014, η μέρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε κατά πόσο είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα αυτής της Σύνοδου Κορυφής. Και φυσικά θα έχουμε και ένα κοινοβούλιο που θα παίξει το ρόλο ατμομηχανής σε αυτή την επιτάχυνση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Θα συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση με τους Ολλανδούς συναδέλφους μας μετά από μια σύντομη ε, διακοπή για να καλωσορίσουμε μετά τους νέους μας καλεσμένους. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Έτσι, με σχετικά ανεπίσημο τρόπο. Να επαναλάβω τους χαιρετισμούς μου και το θερμό καλωσόρισμα προς τους ομολόγους μας από την Βουλή των Αντιπροσώπων των κάτω χωρών. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις ε, δικές σας σκέψεις, ε, τις προτεραιότητές και την προσέγγιση της Ολλανδικής Βουλής σε θέματα άμυνας. Να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια το έργο της υποεπιτροπής μας. Είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάγεται στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο πρόεδρος Σερμαν Μπρόκ θα έρθει σε λίγο. Η δική μας υποεπιτροπή ως βασική της εντολή έχει κατά κάποιο τρόπο ως έργο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι κάπως αδόκιμος όρος, αλλά ε, εποπτεύει τις... Ε, επιχειρήσεις ε, για τις αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Βλέπετε εδώ τον κύριο Πάσκου, τον ε, κύριο Βαμπάλεν, τον Άντριο Ντάφ και τον υποφαινόμενο που ε, τακτικά πηγαίνουμε επιτόπου στις διάφορες επιχειρήσεις της Ένωσης είτε για την καταπολέμηση της πειρατείας, στη Σομαλία, είτε πολιτικού χαρακτήρα στο Κωσυφοπαίδιο ή στη Γεωργία. Πρόσφατα πήγαμε στο Μαλί με τον Ιαν Μπάσκου και στην Ιγυρία και μετά παρακολουθούμε αναφορές από, τους, από τα μέλη των αποστόλων αυτών και έχουμε και κάποιες συζητήσεις που δεν καταλήγουν υποχρεωτικά σε αποφάσεις αλλά αφορούν πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι οι διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου. Και θα θέλαμε να επισυπομπήσουμε και κάποιες προτάσεις μας και το φθινόπωρο στην ετήσια έκθεσή μας θα κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και θέλουμε αυτή η έκθεση να περιλαμβάνει ένα απολογισμό των αποστολών μας και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μας. Επίσης, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ασχολούμαστε και με τον προϋπολογισμό της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, γιατί ο προϋπολογισμός της πολιτικής αυτής είναι ένας προϋπολογισμός που μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί δυνάμει της συναπόφαση συμμετέχουμε στη διαμόρφωση αυτού του προϋπολογισμού. Και τώρα οι πολιτικές αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ΚΕΠΑ είναι όλο και περισσότερος και προϋποθέτουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον ως προς το δημοσιονομικό του σκέλος. Και θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό γιατί το λέω και στις ε, συζητήσεις που έχουμε με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το λέω ως Γάλλος, εγώ δεν γνωρίζω την Ολλανδική Βουλή και δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι οι συνάδελφοι δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των στρατιωτικών και των πολιτικών επιχειρήσεων που γίνονται όλες τα πλαίσια της κοινή ε, πολιτικής άμυνας και πολλές φορές οι εθνικοί βουλευτές δεν γνωρίζουν ότι ε, για τις πολιτικές επιχειρήσεις ε, η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ενώ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξασφαλίζεται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οπότε, από την άποψη της ε, συμμετοχής μας σε τέτοιου επιχειρήσεις και τη συμμετοχή μας στον προϋπολογισμό έχουμε κάποιες ενισχυμένες αρμοδιότητες, κάτι που φαίνεται ότι το αγνοούν οι συνάδελφοι εθνικοί βουλευτές και μερικές φορές επικρίνουν αυτές τις αποστολές. Δεν ξέρω, Άντριο, εσύ που είσαι Βρετανός, αν συμφωνείς, πάντως νομίζω ότι και οι δικοί σου συνάδελφοι και οι Γάλλοι ε, μερικές φορές εξαπολύουν σφοδρές επικρίσεις κατά το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για τη θέση του στα θέματα της ασφάλειας και άμυνας. Η, επιστολή μας, η Επιτροπή μας, η υποεπιτροπή μας παρτίζεται από 32 μέλη, αλλά πολύ σπάνια είμαστε όλοι παρόντες. Το γνωρίζετε αυτό και από τις δικές σας εργασίες. Έχουν πολλές υποχρεώσεις συνάδελφοι. Πάντως έχουμε μερικά μέλη που ε, είναι πολύ επιμελή και πολύ τακτικά στις συνεδριάσεις και πολύ ικανά. Πάντως ο Γιάννη Πάσκου, πρώην ε, για πολλά χρόνια στη Ρουμανία οδήγησε ουσιαστικά την ε, Ρουμανία στο ΝΑΤΟ και έχουμε πολλούς ε, συναδέλφους μέλη της Υποεπιτροπής ε, που είναι βετεράνοι σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και έχουν πάρα πολλές γνώσεις σχετικά. Αυτά ήταν εν λίγα λόγια, μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας και έχετε εσείς το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Ντανζάν, ευχαριστώ για το θερμό σα. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, γιατί υπάρχουν και αρκετοί Ολλανδόφωνοι εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή σας υποδοχή. Η Επιτροπή Αμυντικών Θεμάτων του Ολλανδικού Κοινοβουλίου επισκέφτεται σήμερα τις Βρυξέλλες και κανονίζουμε όλα τα ζητήματα των Βρυξελών, διμερείς επαφές με τους Βέλγους, Ξέρετε πως ε, ίσως κάνουμε κάποια... Έχουμε κάποια κοινά έργα στον τομέα της άμυνας με τους Βέλγους και συναντηθήκαμε και με τον κύριο Πιέρ Λιμόν, τον Γενικό Γραμματέα του... της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που πάντα ενδιαφέρει την Ολλανδία. Οπότε λογικό είναι σήμερα ε, η τελευταία μας συνάντηση να είναι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Άντριο Ντάφ γνωρίζει πως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο για το ότι βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα ε, οι εθνικοί βουλευτές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αδέρφια θα έλεγα, ε, τέσσερις συνάδελφοι είναι εδώ, δύο είναι εδώ πέρα από το φιλελεύθερο κόμμα του κυρίου Φαντάλεν και οι δύο είναι εκπρόσωποι για τα ζητήματα άμυνας ε, του ΒΒΔ και, και η κυρία Άισινγκ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών του Εργατικού Κόμματος και το άλλο κόμμα του συνασπισμού δηλαδή, του κυβερνητικού και τέλος η κυρία Χάτσι ε, των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και οφείλω να πω πως δυστυχώς πρέπει να φύγει μέσα σε 10 λεπτά αλλά κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω λοιπόν πως ε, η στιγμή που ε, συναντιόμαστε είναι πάρα πολύ ευνοϊκή καθώς πλησιάζουμε προετοιμάζουμε το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο του Δεκεμβρίου και όλες οι χώρες μας έχουν στόχο να βελτιωθεί η συνεργασία. Καμιά φορά λέμε πως ε, το μόνο το οποίο είναι κοινό είναι η λιτότητα και το ότι όλοι υποφέρουν στις χώρες όπου ζούμε και προφανώς ε, αυτό επηρεάζει και τους ε, αμυντικούς προπολογισμού και με τα προγράμματα αυτά της λιτότητας έχουμε διάφορα ζητήματα και έτσι προωθείται και η ενισχυμένη συνεργασία και θα θέλαμε βεβαίω να συζητήσουμε μαζί σας το πώς βλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτημα αυτό. Ξέρουμε πως ε, από πλευράς ε, pooling and sharing το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα πιο πρόδευτικα θα έλεγα κοινοβούλια σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε. βεβαίω είναι προφανές πως υπάρχει το ζήτημα της κυριαρχίας, ειδικά σε αυτόν τον τομέα, αλλά νομίζω πως με 180 δισεκατομμύρια ευρώ που ξοδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω πως ε, θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε η μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων μας. Εγώ τώρα δεν θα κάνω κάποιες ε, πολιτικές δηλώσεις, μια που είναι εδώ πέρα όλοι εκπρόσωποι των κομμάτων. Οπότε θα δώσω τον λόγο σε εσά και μπορεί ίσως να ακολουθήσει κάποια συζήτηση για κάποια θέματα τα οποία είναι σημαντικά και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Έλμαρ Μπρόκ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, ε, ήρθε και εκείνο. Σας χαιρετίζω. Ε, γεια σας και από μένα, χαίρομαι που σας βλέπω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγγλικά ή γερμανικά. Yeah. Äh, so versteht man mich schon nicht und wenn es in Französisch ist, schon gar nicht. Ε, τώρα γαλλικά μην τα, μην τα παραλέμε, εντάξει. Χαίρομαι που ήρθατε. Θα ήθελα να κάνω να πω κάποια πράγματα. Ελπίζω εν ώψη της ε, Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου να ενταθούν οι συζητήσεις μας για να έχουμε τελικά μια ένδειξη για το με ποια βάση πρέπει να κινηθούμε και να συζητήσουμε τον Δεκέμβρη. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που απαιτούν πολιτική βούληση. Έχουμε την απόφαση της Δευτέρας που μας πέρασε του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και αφορούσε την εξαγωγή όπλων και de facto μιλάμε για μια επανεθνικοποίηση αυτού του θέματος μετά το γαλλικό και το βρετανικό βέτο. Και από ό,τι φαίνεται η αντίδραση της Ρωσίας μας οδηγεί στο ότι έχουμε ένα άλωθι για να πούμε πως μπορούμε να στείλουμε και να εξαγάγουμε, εννοώ μαχητικά αεροπλάνα στη Συρία. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, ε, γιατί πρέπει ε, να έχουμε και μια φωνή η οποία θα ακούγεται, να μην είμαστε συνεχώς διχασμένοι. Και ακόμα και τα εθνικά κράτη πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτές τις δυνατότητες επιρροής, γιατί η επιρροή της ε, Ευρώπης οφείλεται στην ενότητα εάν υπάρχει. Και φοβάμαι πως αυτό δεν το συνειδητοποιούν συχνά ούτε η δική μου κυβέρνηση, ούτε άλλες. Έχουμε το θέμα της δομημένης συνεργασίας, το τι θα γίνει από εδώ και μπρος, πώς θα χρηματοδοτηθεί και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο θέμα των προμηθειών. στη Γερμανία είχαμε ε, τελευταία κάποιες εξελίξεις σε σχέση με την υπηρεσία ε, προμηθειών. Ε, αλλά βλέπετε πως εμείς μπορεί να θέλουμε κάποια πράγματα, αλλά οι υπάλληλοι εκεί πέρα που κάθονται στις θέσεις δεν αλλάζουν μυαλά, επιμένουν και όλο αυτό τελικά κοστίζει και εγώ θεωρώ πως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη κατανομή εργασίας όσον αφορά τον τομέα της αμυντικής πολιτικής και ε, των προμηθειών. Και εκεί πέρα νομίζω πως ε, πρέπει να δούμε και το τι γίνεται και με τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβουλία. Ενδιαφέρον όμως θα ήταν να μας πείτε εσείς από την Ολλανδική Σκοπιά πώς τα βλέπετε αυτά, πολυμερείς, διμερείς συνεργασίες. Εγώ είμαι από την Βεσφαλία, ξέρετε, και ξέρω εκεί πέρα πως υπάρχει στενή συνεργασία Ολλανδικού και Γερμανικού στρατού ναι, κάτι το οποίο βεβαίως ε, βρίσκω υπέροχο αλλά νομίζω πρέπει να συνεχιστεί ειδικά βλέπω πως υπάρχουν ε, προβλήματα από τη γερμανική πλευρά με την ε, κοινοβουλευτική επιφύλαξη που υπάρχει πάντα από πλευράς Γερμανίας για οποιαδήποτε επιχείρηση και έτσι δυσκολεύουν τα πράγματα θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και τη δικιά σας εμπειρία για τα προβλήματα της ε, συνεργασίας. Υπάρχει και το γνωστό Eurocore, η γαλλογερμανική ε, μεραρχία ε, και άλλες συνεργασίες και η Πολωνία συνεργάζεται με άλλες χώρες και οπότε πρέπει να υπάρξει μια κοινή επιχειρησιακή συνεργασία. Γι' αυτό χαίρομαι για το ότι έχουμε τη δυνατότητα για αυτές τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, άλμαρα. Γιάννου Πάσκου είχε ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν μιλάμε για συγκέντρωση και κοινή χρήση ικανοτήτων, αυτό σημαίνει βασικά κατ' ουσίαν ότι ε, τα στατεύματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Οι δύο χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιούν ναι για την χρήση. Ε, και άρα θα κληθούν τα δύο κοινοβούλια να πούν ναι. Και ως προς αυτό πιστεύω πως γνωρίζετε πως ε, η ενίσχυση διμερών ή τριμερών συνεργασιών ανάλογα με τη μορφή της κοινή χρήσης ε, θα πρέπει να προέλθει από το κοινοβούλιο, θα πρέπει να γίνεται στο επίπεδο του, των κοινοβουλίων. Αν μιλάμε για μάχη με σωμάδες, για χρήση αυτών ε, και έχουμε τρεις χώρες που συμμετέχουν, τα κοινοβούλια των τριών χωρών θα πρέπει να πούν ναι Άρα λοιπόν, ως προς αυτό, θα πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο πέρα από τη σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά. Τα Εθνικά Κοινοβούλια τα ίδια μεταξύ τους. Ανάλογα με το είδος της ε, κοινή χρήσης που έχουν, θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Θα, πρέπει να, θα, ήθελα να έχω τη γνώμη σας. Ας πούμε με τους, ε, το Βέλγιο έχετε ισχυρότερη συνεργασία από ό,τι με άλλες χώρες όπου δεν έχετε πολύ sharing. Ο Άντριου. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να πω πόσο καλό είναι που βρίσκεστε εδώ. Νομίζω πως χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερο διάλογο ανάμεσα στις επιτροπές αμήνης των ε, κοινοβουλίων. Και ζητώ συγγνώμη γιατί θα πρέπει να αναχωρήσω σε δύο λεπτά. μάλλον κατά τις 6. Θέλω όμως να σας ρωτήσω για την απόφαση του Συμβουλίου να, να καταργήσει το εμπάργκο όπλων. Ποια είναι η θέση Ε, ήρθε σε επαφή ο Υπουργός Αμήνης σας, μαζί σας. Και τι θα κάνετε τώρα που λήφθη η απόφαση. για να παρακολουθήσετε τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως θα προσπαθήσω να μοιράσω τις ερωτήσεις και μάλλον τις απαντήσεις ανάμεσα στα διάφορα μέρη. Τώρα για τη κρίση της Συρίας θα απαντήσω εγώ. Ο Έλμαρ Μπρόκα αναφέρθηκε στη συνεργασία με τη Γερμανία και το γερμανικό Parlaments Vorbehalt. Διαδικαστικά έχουμε κάτι παρόμοιο. Και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Έσινγκ που ασχολείται με αυτή τη διαδικασία και την έχει ήδη κάνει μια-δυο φορές να απαντήσει. Ίσως θα μπορούσε επίσης να πει δύο λόγια και για το πρόσφατο Memorandum of Understanding που υπέγραψαν οι υπουργοί μας ε, μήνες πριν από μια εβδομάδα καθώς και την ανάπτυξη των Patriot στην Τουρκία. γιατί τμήμα του Εμμογιού αφορούσε το πυράβλους Patriot. Και έπειτα να ζητήσω από τον κύριο Φάικ ίσως να πει δύο λόγια όσον αφορά την κοινή χρήση mutualization of assets, την κοινή χρήση των ικανοτήτων, που στην ουσία είναι άλλα λόγια για να πούμε pooling and sharing. και για το βελγικό παράδειγμα και για το τι κάνουμε μαζί να θα ζητήσω από την κυρία Μπέρξεν να απαντήσει. Μου επιτρέπετε? Κυρία Άσλη, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μας εδώ. Μικροφωνή στο μικρόφωνο δυστυχώς. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα και χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Βαμπάλεν που είναι παλιός γνώριμος της Ολλανδικής Βουλής είναι ακόμη στην αίθουσα. Είναι μαζί μας. Ακόμη ο κύριος Βαμπάλεν και με ιδιαίτερη χαρά τον ξανασυναντούμε. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Συζητήσαμε σήμερα με κάποιους συναδέλφους από τη Βελική Βουλή ε, τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε ώστε να περάσουμε από τις συναντήσεις στις αποστολές γιατί μερικές φορές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες εξαιτίας και του συντάγματος. Το συντάγμα προβλέπει ότι δεν χρειάζεται να ενημερώνεται το κοινοβούλιο από την κυβέρνηση ή μάλλον ενημερώνεται αλλά δεν χρειάζεται να δώσει και την έγκρισή του. Στη Γερμανία ισχύει κάτι διαφορετικό. Αυτό οφείλεται στην ιστορία της Γερμανίας, σε μακροχρόνιες συζητήσεις που είχατε στη Γερμανία, στο σύνταγμά σας, και συζητήσαμε πολύ εντατικά το θέμα αυτό και τις διαδικασίες με τους Βέλγους ομολόγους μας. Και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ντεμπρούκε, είπε γιατί δεν προσπαθούμε με μερικές χώρες να εξακριβώσουμε τις διαδικασίες που ισχύουν για τις διάφορες αποστολές και εκθέσεις για τις αποστολές, γιατί στην, στην Ολλανδία έχουμε 11 κόμματα στη Βουλή μας. 11 κόμματα. Δεν είναι εύκολη συνεννόηση. Οπότε η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα μέχρι να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Στο Βέλγιο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στο Βέλγιο πήραν αμέσως την απόφαση για τη Λιβύη. Δύο τρίτα όμως ε, ε, του Κοινοβουλίου συμμετέχει στο κυβερνητικό συνασπισμό, οπότε είναι πολύ διαφορετική διαδικασία. Απαντώντας λοιπόν σε ερωτήσεις σας κύριοι Μπροκ και Πάσκου, το πιο σημαντικό είναι ο διάλογος μεταξύ των κοινοβουλίων. Και ξεκινήσαμε αυτό το διάλογο σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις με τους Βέλγους ομολόγους μας τον Οκτώβριο. Και το Συμβούλιο, η Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες δηλώσεις, κάθε βουλή χωριστά, αλλά και κάποιες κοινέ δηλώσεις των κοινοβουλίων. Γιατί το pooling and sharing και smart defense, smart buy, όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει πολλές φορές. Χρόνια ολόκληρα τα ακούμε. Οπότε θα πρέπει να συνδυάσουμε όλα αυτά τα θέματα και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα αυτό. Αλλά για σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτά. Α, για το μνημόνιο συνεννόησης. Ναι, σωστά το επισημάνατε. Την περασμένη ο υπουργό Άμυνα μας ε, υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεννόησης για τέσσερα προγράμματα με την Γερμανία. Πάτριο της Τουρκία, υποβρύχια, στενή συνεργασία στο, στο Μίνστερ. Θα το ξέρετε αυτό. Έχουμε κοινά σχέδια με πολλές χώρες, αλλά και διμερός και πολυμερός έχουμε ακόμη πολύ έργο μπροστά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα. Είχαμε πολλές ε, συζητήσεις σήμερα και για την πρώτη γερμανική στρατιά και τους σχηματισμούς μάχης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχηματισμοί αυτοί δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Και αναζητούμε κάποια λύση γιατί πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ή αυτά χάνονται, ξέρετε, άμα τα αφήσει αφήνουν. Έχουμε θέμα βεβαίως εθνικής κυριαρχίας και πολυπλοκότητας πολιτικής. Η πολιτική πολυπλοκότητα, παραδείγματος χάρη, αυξάνεται όταν ε, συμμετέχουν περισσότερα κράτη στη χρήση των μέσων το γαλλογερμανικό σώμα έχει, το, συγχωρείτε, ολλανδογερμανικό σώμα έχει δύο χώρες μόνο και δύο κοινοβούλια εμπλέκονται και είναι ευκολότερο από α, ε, το να εμπλέκονται τα 27 κρατημέλη. Αλλά τίθεται το ζήτημα του μέλλοντος των σχηματισμών μάχης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει βέβαια και το ζήτημα στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την πολιτική, αλλά έχουμε και μια άποψη εδώ πέρα. Εμεί θεωρούμε πω οι σχηματισμοί μάχη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να απαντήσουν σε τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, το κόστος. Ποιο πληρώνει για τη χρήση των μέσων, εάν υπάρχει ανάπτυξη αυτών των σχηματισμών θα είναι προς το συμφέρον και των 27 κρατών μελών. Οπότε, ποιος πληρώνει. Δεύτερον, τι είναι αυτοί οι σχηματισμοί. Είναι μόνο κατά ξηρά ή κατά αέρα και θάλασσα. Επίσης, ευελιξία. Μπορούμε να εργαστούμε και ε, με στοιχεία ε, του κάθε σχηματισμού ή ολόκληρο το σχηματισμό υποχρεωτικά. Και τέλος θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σχηματισμή γιατί μαθαίνουμε κάποια πράγματα, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε ως χώρες, ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ζήτημα είναι, το ερώτημα είναι ε, το εάν επαρκεί αυτο και το συζητάμε αυτό και στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Για το τελευταίο θέμα, για τις διμερείς επαφές ε, με τους Βέλγους, η κυρία Μπέργμους ίσως μπορεί να μας πει κάποια πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για άμυνα, οι πολιτικοί ε, ασχολούνται με το γιατί και το τι κάνουμε κάτι. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ ως πολιτικός είναι πως στρατιωτικοί μας σχηματισμοί ε, ήδη ασχολούνται με το πώς και το κάνουν. Ε, οπότε κάποια πράγματα συμβαίνουν ήδη και εμείς οι πολιτικοί ακόμα συζητάμε το πώς θα γίνουν. Ενώ τα πράγματα συμβαίνουν και εμείς ψάχνουμε τους κανόνες μεταξύ κοινοβουλίων κτλ. Και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό. παράδειγμα από την περιοχή που μένω εγώ, στο Den κοντά, εκεί πέρα συνεργαζόμαστε με, γιατί είναι κοντά ο ναύσταθμος εκεί πέρα και συνεργάζονται με το βελγικό ναυτικό και τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Εγώ έχω βέλγους γείτονες ε, που εργάζονται Και Ολλανδοί πήγανε στην στο Βέλγικο ναύσταθμο, για τρία χρόνια. Οπότε η συνεργασία πάει μια χαρά, σε κάθε επίπεδο. Και το θέμα είναι απλά να γίνει κάτι. Έτσι, λιγότερα λόγια και να περάσουμε στις πράξεις. Put aside, perhaps, ε, Πρέπει να αφήσουμε τα πολλά τα λόγια και να περάσουμε στις πράξεις. Να μας τα πει κυρία Δηλαδή αναλύουμε το τι γίνεται σε κάθε χώρα και βεβαίω μετά προχωράμε συνεργασία. Αλλά το καλό είναι ότι αυτά τα πράγματα ήδη συμβαίνουν. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ιδιαίτερα σε ό,τι φορά το πολεμικό ναυτικό έχουμε ε, συνδυασμένες και προσπάθειες και ε, δομή διοίκησης με το βελγικό ναυτικό είναι πραγματικά η πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της ε, συνεργασίας σε ό,τι αφορά το πολεμικό ναυτικό. Ε, Άντριου Ντάφ, ρωτήσατε για τη Συρία. Ε, στο δικό μας κοινοβούλιο δεν είναι ο Υπουργός Άμυνας αυτός που μας ενημερώνει, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυτός είναι αρμόδιος. Και φυσικά δυσανασχετήσαμε με την απόφαση αυτή. Αυτή ήταν αυτό το, το, το κυρίαρχο αίσθημα στην Ολλανδική Βουλή. Δυσαρεστηθήκαμε με την άρση του εμπάργου προς τη Συρία γιατί έχουμε 72 ψηφίσματα σχετικά και είδαμε ότι οι Ρώσοι έλαβαν αυτή την ατυχή απόφαση ε, και τη χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα για να συνεχίσουν να, ε, πουλάνε, και παραδίδουν όλο και περισσότερα όπλα πολύ περισσότερα από ό,τι προηγουμένως. Και ήδη είχαν το πράσινο φως από την ε, Συριακή Αντιπροσωπεία για μετάβαση στη Γενέβη για διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει παραμείνει μεγάλο περιθώριο λιμών. ούτε για αυτούς ούτε για την αντιπολίτευση που αρχίζει και διαλύεται. Και τη στιγμή που είδαμε το εμπάργο των όπλων, ακούσαμε την ομιλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον αρμόδιο στρατηγό που είπε ότι δεν έχει πια τον έλεγχο των στρατευμάτων και δυστυχώς πολύ αργά και κατόπιν εορτής δράσαμε και μάλιστα με πολύ μικρές ευέλειες προσπάθειες και πριν από ένα χρόνο η, μετα... Η μεταφορά της εξουσίας ήταν τμήμα των συμπερασμάτων και μάλιστα συμφωνούσαν σε αυτή τη μεταφορά εξουσίας και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Και ένα χρόνο μετά έχουμε διαπιστώσει τη σύγχυση και το τεράστιο χάος που επικρατεί στη Συρία. Και πολλοί Σύριοι δεν αναφέρουν, δεν αυτοχαρακτηρίζονται καν ως Σύριοι, αλλά με βάση την, το που ανήκουν θρησκευτικά έχει δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα μεταξύ των διαφόρων αρέσεων και δογμάτων και ε, έχουμε και την κατάσταση στο Ιράκ, πολλές ανησυχίες για το τι συμβαίνει στην Ιορδανία. Και ούτως ή άλλως το εμπαργό των όπλων έχει αρθεί de facto. Και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είπαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν παραδόσεις όπλων πριν την 1η Αυγούστου. Θα δούμε τελικά τι θα συμβεί. Εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο για τη δεύτερη συνάντηση της Γενέβης. Δεν πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ειρηνευτική συμφωνία αν κανένα από τα μέρη δεν πιστεύει ότι μπορεί να κατάγει στρατιωτική νίκη. Και αν δεν θεωρούν ότι μπορούν να νικήσουν στρατιωτικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα για ειρηνευτική συμφωνία ή για περιφερειακή εκεχηρία για κατάβαυση του πυρός. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόφαση αυτή έχασε οποιαδήποτε δυνατότητα επιρροής ε, έχει στην κατάσταση. Η, γνω... η αυτή η άποψη ε, βρίσκει πολλούς υποστηρικτές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, παρόλο που δεν είχαμε επίσημες ε, ε, αποφάσεις και συγκεκριμένη οριστική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο αλλά το ακούσαμε και από τον αρμόδιο υπουργό άμυνα τη Γαλλία, τον κύριο Βημό, που έκανε αντίστοιχα σχόλια την περισμένη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τις μάχημες ομάδες στην ετήσια μας έκθεση εκφράζουμε τη θλίψη μας για το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ αυτές οι μάχημες ομάδες. Και μερικοί λένε κοιτάξτε τους ε, μιλιταριστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλουν πάση θυσία να χρησιμοποιήσουν τις μάχημες ομάδες ενώ αν τις χρησιμοποιούμε σημαίνει ότι δεν υπάρχει κρίση Άρα γι' αυτό δεν χρειάζονται οι μάχοι με ομάδε. Ενώ εμεί λέμε ότι κρίμα που δεν χρησιμοποιούνται εκεί που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί. Θέλουμε περισσότερη ελαστικότητα και ευελιξία στη διαδικασία για την ενεργοποίηση και χρήση αυτών των ε, μάχημων ομάδων. Γιατί πίσω από τις μάχημες ομάδες ουσιαστικά κρύβεται το πραγματικό πρόβλημα. Μερικές φορές ε, το δέντρο μας κρύβει ολόκληρο το δάσος και ουσιαστικά το θέμα των μάχημων ομάδων είναι περιθωριακό σε σχέση με το συστικό πρόβλημα που είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης των χωρών να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά εργαλεία σε μια κοινή πολιτική. Το διαπιστώσαμε αυτό με τη Λιβύη, με το Μαλί. Υπάρχει μεγάλη απροθυμία και πολλές επιφυλάξεις των κρατών μελών. Για να μην πω εχθρότητα από κάποια κρατημέλη, τουλάχιστον ε, μεγάλη αντίσταση προθυμία των κρατών μελών να εξετάσουν ε, ως πιθανή φυσική ε, διέξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρήση ε, στρατιωτικής δύναμης. Και το συζητήσαμε αυτό και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Διαπιστώνουμε ότι ε, πριτανεύουν οι πολιτικές λύσεις και η υπηαδύναμη δεν αμφισβητούμε αυτή την πολιτική και είναι προς την της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τέτοια φιλόδοξη πολιτική για τις πολιτικές αποστολές και την ήπια δύναμη, το soft power. Αλλά κρούμε πολύ τακτικά το κόδωνα του κινδύνου στην υποεπιτροπή μας. Ότι το στρατιωτικό σκέλος ναι μεν είναι περιθωριακό και είναι ίστατη λύση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραμελείται. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καυχέται ότι υιοθετεί μια σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν νοείται χωρίς στρατιωτικό σκέλος. Οπότε, οι μάχημες ομάδες αποτελούν και ένα σημαντικό σύμβολο. Δεν είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε, αλλά πολύ φοβούμαι ότι πίσω αυτή τη συζήτηση για τις μάχημες ομάδες κρύβεται μια πολύ πιο σημαντική και θεμελιώδης συζήτηση για την πολιτική βούληση των κρατών μελών να προσφύγουν σε τέτοια μέσα αλλά και την έλλειψη βούληση στις ε, ευρωπαϊκές δομές, γιατί είχαμε και την συζήτηση για την κρίση στη Λιβύη και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε σφοδρή κριτική για την έλλειψη σχεδιασμού και πρόληψης ε, που χαρακτηρίζει μερικές φορές τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και οι ίδιες επικρίσεις θα μπορούσαν να σκεφτούν και στην περίπτωση του Μαλή. Πολλές φορές ε, Επισημάναμε εδώ ότι δυστυχώς οι πολιτικές ασφάλειες και οι αναπτυξιακές πολιτικές στο Σαχέλ ε, δεν θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένες, αλλά θα πρέπει να είναι αλληλένδετες. Και ότι το τμήμα της ασφάλειας δυστυχώς ε, υστέρησε σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτό είναι μια δυναμία των πολιτικών μας και των θεσμικών μας οργάνων. Και δυστυχώς ε, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό ο συντονισμό μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, που είναι σχετικά νεοπαγή, οπότε είναι, ε, ε, χρειάζεται κάποιο χρόνο για να λειτουργήσει πλήρω, μεταξύ αυτή τη ΕΕ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και υπάρχει καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Και μάλιστα η έλλειψη συντονισμού μεταξύ αυτών των δύο θεσμικών οργάνων μα. Ε, γυρίζει πολύ πίσω και δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις στο σχεδιασμό και στην πρόληψη, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα σε σημαντικές αποφάσεις και σε σημαντικές περιστάσεις. Και αυτές οι επικρίσεις είναι απόλυτα τεκμηριωμένες. Δεν είναι καθόλου επιπόλες. Ούτε θέλουμε συστηματικά να επιρρύπτουμε την ευθύνη στα θεσμικά όργανα. Γιατί θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να είναι κυρίαρχα και το διεκδικούν αυτό συνεχώς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αποποιούνται των ευθυνών τους. Αλλά υπάρχουν και θέματα που μπορούμε να τα βελτιώσουμε σε επίπεδο Βρυξελών και κυρίως τη διάρθρωση μεταξύ των διαφόρων θετικών οργάνων. Για να δώσουμε πιο αποτελεσματικές και πιο άμεσες αντιδράσεις ε, σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Με το Γιάν Πάσκου όταν πήγαμε στον Νίγηρα πρόσφατα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια πολιτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί μείναμε ευρώντιτοι από τις δυσκολίες που έχουν σε επίπεδο επιμελητίας, σε επίπεδο υλικό, ε, για την ανάπτυξη αυτών των αποστολών και την εφαρμογή τους. Και οι αποστολές αυτές είναι πολύ χρήσιμες, γιατί υπάρχει μεγάλη απόπειρα και απειλή για αποσταθεροποίηση εξαιτία τρομοκρατίας στο Σαχέλ. Και μάλιστα πολλές φορές οι συνθήκες για τις αποστολές αυτές είναι απαράδεκτες. Φαίνεται ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως ε, τις δυνατότητες της συνθήκης της Λισαβόνας. Οι πολιτικές μας αποστολές σήμερα, το 2003, τη σήμερα ημέρα, είναι οι ίδιες με αυτές που είχαμε το 2003, 2004 και 2005 όταν αυτές οι πολιτικές αποστολές βρίσκονταν ακόμη στα σπάργανα. Δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε την αυτοκριτική και στις Βρυξέλλες, χωρίς φυσικά να παραμελούμε τις ευθύνες για των κρατών μελών. Ο κύριος Βανμπάλεν. Ευχαριστώ κύριε Ντανζόν. Έχω μία ερώτηση προς την Ολλανδική Αντιπροσωπεία και αφορά τις δυνατότητες. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν δυνατότητες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ολλανδία για τον διάδοχο του F-16, του μαχητικού. Δεν θέλω τώρα να μπω εγώ σε μια εθνική συζήτηση, αλλά η Ολλανδία, ό,τι και αν επιλέξει, θα αγοράσει ένα διάδοχο του F-16, γιατί χωρίς δυνατότητες ε, δεν γίνεται τίποτα. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν ε, την άποψη των σοσιαλδημοκρατών και των φιλελευθέρων. Κύριε Φαντάλ, σας ευχαριστώ για την ουδέτερη ερώτησή σας και την πρότασή σας που θέλετε να ακούσετε και τους δύο κυβερνητικούς εταίρους, αλλά μπορώ να σας πω ήδη πως η Ολλανδία ήδη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αποφάσιζε πως όταν, όπου έχουμε στρατεύματα σε άλλη χώρα θέλουμε να βασιζόμαστε σε δική μας αεροπορική υποστήριξη. Και... Κυρία Άισιγγεν και κύριε Φάλκ, μια που και οι δύο ασχολείστε με αυτό το θέμα μπορείτε να διαφορτήσετε τον κύριο Φαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι αν θα αγοράσουμε διάδοχο του F-16. Η απάντηση είναι ναι ξεκάθαρα. Δεν θα αναφέρω τώρα το, τον κλάδο. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, όπως είπε ο κ. Σοντάλμ. Και εμένα η απάντησή μου είναι η ίδια. Δεν θα έχουμε στρατεύματα χωρίς ε, μαχητικό αεροσκάφος. Χρειάζεται αεροπορική υπεροχή και ιστορικά έχει ε, αποδειχθεί πως χρειάζεται και μαχητικά αεροσκάφη. Χρειάζεται και άρβιλο βεβαίως επιτόπου να πατήσει, αλλά χρειάζεται και μαχητικό αεροσκάφος. Οπότε θα υπάρξει διάδοχος. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η αεροπορία μας είναι ακόμα στο Αφγανιστάν, έτσι από το αεροδρόμιο του Μαζάρι Σαρίφ επιχειρεί και παρέχει εγγύηση εκεί υποστήριξη στις μαχικές δυνάμεις. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής μπορώ να σας δείσω τη γνώμη σα για την αντίληψη στο, Ευρω... Ολλανδικό Κοινοβούλιο για τις αποστολές πολιτικού και στρατικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι αποστολές ε, παρακολουθούνται στενά, γιατί και εδώ θα πρέπει να πω ότι γνωρίζω ορισμένα εθνικά κοινοβούλια που έχουν μια εικόνα αρκετά μακρινή, απόμακρη των αποστολών και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται στο Ολλανδικό επίπεδο γνωρίζοντας ότι στο Συμβούλιο στο τέλος του έτους ε, θα προσεγγιστούν ε, τρία μεγάλα, μεγάλα θέματα και το πρώτο είναι οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν ήδη κάποιες θέσεις που διαγράφονται στο Κοινοβούλιο, το Ολλανδικό. Ναι. Κατά τη διάρκεια των ετών, κατά τη διάρκεια των αποστολών στις οποίες συμμετείχαν οι κατοχώρες, αναπτύξαμε μια αρκετά γνωστή δομή και για τις πολιτικού χαρακτήρα και για τους στρατιωτικού χαρακτήρα αποστολές. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση. Η αποστολή μας στο Αφγανιστάν εντό της ΙΣΑΦ ήταν ε, τμήμα ε, πολιτικής αποστολής. Ήμασταν τμήμα του ΣΥΜΙΚ, δηλαδή ε, επιχειρήσει στρατιωτικού και πολιτικού χαρακτήρα. Συμμετείχαμε στις δράσεις εκπαίδευσης των, των αποστολών εκεί. Τα γνωρίζετε, γιατί ήταν διαφορετική φύση αποστολή από ό,τι είχαμε παλιότερα. Πρόκειται για μια καθολική προσέγγιση, για μια τρισδιάστατη μεταξύ μας, λέμε, προσέγγιση, δηλαδή άμυνα, ε, επιχειρήσεις και ανάπτυξη. Το έχουμε συζητήσει, ε, το συζητήσει μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας μας, αναφέρθηκε και ο κύριος Βανμπάλεν συμμετείχε μάλιστα σε αυτή την, την, την ιδέα που είχαμε μέσω μιας έκθεσης με τον κύριο Βανμπάλεν και τον κύριο Κούντρες ε, και στη σχέση με τον ΝΑΤΟ, κάποιοι από εσάς θα τους γνωρίζετε. Πάντως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των αποστολών μας και από τη δική μας πλευρά του εργατικού κόμματος πάντοτε λέμε ότι καταρχήν συμμετέχουμε στις υποστολές πολιτικής φύσης, δηλαδή πρώτα διπλωματία και ανάπτυξη και αν χρειαστεί και το στρατιωτικό τμήμα βέβαια. Δεν θα διστάσουμε αν χρειαστεί. Πάντως καταρχήν ε, θέλουμε την πολιτική διάσταση. Και Επίσης ήταν πολύ σημαντικό να συζητήσουμε την αποστολή ΣΥΜΕΚ που και εδώ συζητήθηκε πολύ νομίζω. Για άλλου είδους αποστολές πάλι εξετάζουμε την ε, τρισδιάστατη προσέγγιση, η καθολική προσέγγιση που είναι πολύ σημαντική για μας. Ένα-δύο πράγματα που και σήμερα συζητήσαμε, συζητήσαμε και το EUTM γιατί είναι ε, πολύ επίκαιρο θέμα. Οι κάτω χώρες δίνουν ε, εκπαιδευτές στην EUTM στην Σομαλία. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή συζητά αν θα πρέπει να συμβάλλει και στο Μαλί. Πάντως ποια είναι η κατάσταση για τις κάτω Οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι στο Κούντους, η εκπαίδευση της αστυνομίας με αρχηγό την Γερμανία στην βόρεια επαρχία του Κούντου. Έχουμε αναπτύξει εκεί στα Άδανα, επίσης, στρατιωτικές δυνάμεις Patriot, πυράβλους Patriot, μαζί με τους Αμερικανούς, καθώς και πολιτικές δυνάμεις και σύντομα θα είμαστε εμείς το αρχηγό, κράτος αρχηγός στην Αταλάντα. Την επιχείρηση Αταλάντα. Αυτές είναι οι βασικές μας επιχειρήσεις. Έχουμε περίπου χίλιους στρατιώτες στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Είχαμε και εδώ ένα καταπληκτικό απολογισμό των δύο αποστολών AUTM πριν μεταβού μάλιστα στη Σο... Σομαλία, όταν ήταν ακόμη στην Ουγγάντα. Πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή, με σχετικά μικρό κόστος και μεγάλο πολιτικό όφελος για το στρατηγικό αυτό τμήμα της Αφρικής. Και ήταν πολύ καλό το έργο αυτών των αποστολών και μάλιστα ε, έδωσαν πολύ μεγαλύτερη προβολή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι το σχετικά μικρό κόστος που είχαν. Και τώρα ε, είδαμε ότι η προέλαση του Σομαλικού στρατού ήταν αρκετά εντυπωσιακή, παρόλο που έχουμε πολύ έργο ακόμη μπροστά μας και έχουμε τακτικές επαφές ε, με την ΕΕΔ το κέρας της Αφρικής και ο ειδικό εκπρόσωπος έρχεται πολύ τακτικά στην Υποεπιτροπή και δίνει έμφαση στην προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση και την εδραίωση των ε, δομών ασφάλειας στη Σομαλία, ε, κατά κύριο λόγο στο στρατό. Και στο Μαλί συναντηθήκαμε με τον στρατηγό Λεκουάντρ, και εκεί γίνεται τεράστιο έργο από την αποστολή, κάτι που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε στην αρχή, γιατί θα πρέπει να αναδιαρθωθεί άρδιν ο στρατός του Μαλή και μάλιστα σε πολύ δύσκολο πλαίσιο και καιρό. Πάντως ε, τα ανώτατα στελέχη της αποστολής UTM έχουν πραγματικά μεγάλες γνώσεις και δεξιότητες, γνωρίζουν καλά την κατάσταση και νομίζω ότι αυτή η αποστολή είναι πολλά υποσχόμενη. Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα γιατί οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιορίστηκαν στις δυνάμεις ε, για την προστασία της αποστολής παρά στο ίδιο το έργο της αποστολής. Κατά τη γνώμη μου αυτό ε, είναι λυπηρό, γιατί όπως μας επιβεώσαν και επιτό αναλύσεις, ο κίνδυνος, μια και βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη, το Μαλί βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και εκεί που γίνεται η ανάπτυξη της αποστολής ε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλε οι απειλέ. Γιατί εντάξει, υπάρχει παντού η πιθανότητα τρομοκρατική απειλή, αλλά ακόμη και στι Βρυξέλλε. Δεν νομίζω ότι ε, ήταν τόσο σημαντική η συμπληρωματική αποστολή προστασία για να εξασφαλιστεί η προστασία της αποστολής αυτή, Νομίζω ότι εκεί κολλήσαμε και χρονοτριβήσαμε πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτή την ε, υποστηρικτική δύναμη προστασίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει συστηματικά να ασκούμε κριτική σε αυτή την κολυσιεργία και τη βραδύτητα στην αντίδραση, που μερικέ φορέ αφισβητεί και την ίδια τη χρησιμότητα τέτοιων αποστολών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, οι αποστολέ EUTM ε, λειτουργούν πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Αταλάντη, και αυτή η επιχείρηση είχε πραγματικά συμβολικό χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν πραγματικά επιθετική αποστολή, επιχείρηση με πολύ καλά αποτελέσματα και ε, και εμείς είδαμε η τα, το έργο αυτής της αποστολής και τη συνεργασία με τους εταίρους και το ΝΑΤΟ. Πάντως το ενδιαφέρον στην επιχείρηση Αταλάντη ήταν οι εταιρικές σχέσεις και με τις τρίτες χώρες. Με τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία με όλες αυτές τις χώρες που ενδιαφέρονται για την ε, θαλάσσια ασφάλεια. Και σίγουρα εκεί υπάρχει μεγάλο έδαφος για εξερεύνηση και για την PSDC, ε, που είναι όχι μόνο απλώς μια προβολή των ευρωπαϊκών ε, μέσων και δυνατοτήτων, αλλά γνήσεις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες, για τις οποίες θα είναι δύσκολος ο διάλογος για την άμυνα, αλλά μπορούμε σίγουρα να βρούμε κοινό έδαφος και κοινό παρανομαστή για την περιοχή του κέρατος της Αφρικής και ενδεχομένω ε, και για άλλες θαλάσσιες περιοχές. Και νομίζω ότι αυτές οι τρεις αποστολές και επιχειρήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και για αυτές τουλάχιστον εξασφαλίσαμε μία παρακολούθηση, εκ του παρακολούθηση και τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Και φυσικά είμαστε πιο αυστηροί με το χαρακτηρισμό των πολιτικών ε, αποστολών. Κάτι που είναι παράδοξο, γιατί οι πολιτικές αποστολές είναι και η καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η οργάνωση μερικές φορές εκεί χωλαίνει. Γι' αυτό και είμαστε πιο επικριτικοί απέναντι σε αυτές τις πολιτικές αποστολές. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόβλημα με την ανάπτυξη αυτών των ε, πολιτικών αποστολών και την, κυρίως την έναρξη, την, έναρξή τους. Και αυτή η βραδύτητα ακριβώς ε, προβάλλει τις αδυναμίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη γραφειοκρατία, την ε, νοθρότητα μερικές φορές των δομών και μεγάλη απώλεια ενέργειας ε, στη φάση της ανάπτυξης και της εφαρμογής αυτών των πολιτικών αποστολών. Δίκιο έχετε κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως από τη δική μας την πλευρά μπορούμε να πούμε πως αν συγκρίνεται π.χ. Ε, τις επιχειρήσεις κατά της πειρατείας στην Αταλάντα με την Ocean Shield του ΝΑΤΟ εμείς είμαστε πιο ικανοποιημένοι με την πρώτη. Είναι μια στρατιωτική επιχείρηση και είναι πολύ πιο αποτελεσματική η ευρωπαϊκή επιχείρηση από την Ocean Shield για τους γνωστούς λόγους. Οπότε, καλό είναι να το λέμε και αυτό που και που. Πως καμιά φορά και η Ευρώπη κάτι μπορεί να κάνει. Έτσι για αλλαγή. Αλλά συμφωνούμε όλοι πως η πειρατεία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο στη θάλασσα. Οι αιτίε βρίσκονται στην ξηρά. Και εκεί πέρα ακριβώς βρίσκεται ε, και εκεί πέρα κολλάει η εκπαιδευτική αποστολή. Τώρα για το Μαλή δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, το εξετάζουμε ακόμα και για την, ε, την εκπαιδευτική αποστολή στη Σομαλία συμμετέχουμε σε όλες τις πτυχές και τις πολιτικές της εκπαίδευσης των δικαστών ε, του κράτους δικαίου κτλ. Εγώ θα ήθελα ε, και η Επιτροπή μου να σας απευθύνει μερικές ερωτήσεις, αν συμφωνείτε. Ε, οι τρεις συνάδελφοι εδώ πέρα. Ποιος θα κάνει τις ερωτήσεις. Έλα, θάρρος. Το πρώτο, η πρώτη μου ερώτηση αφορά τις, ε, τους σχηματισμούς μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως εξής. Ποιες άλλες ευκαιρίες βλέπετε. Συζητήσαμε την ε, Ολλανδογερμανική συνεργασία. Βλέπουμε επίσης συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου και υπάρχει και συνεργασία γαλλογερμανική και συνεργασία από κάτι προς τα πάνω. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Κοιτάξτε, η εντύπωση γενική των μελών αυτής της υποεπιτροπής και των μεταβαστικών πολιτικών ομάδων θα έλεγα πως είναι ότι είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι από τα κράτη-μέλη. Θα θέλαμε ιδανικά να δούμε αυτήν την συνεργασία όσο γίνεται πιο ζωντανή και να προχωρήσουμε αν είναι δυνατόν Έγινε λόγο για bottom-up, αλλά ίσω και top-down. Θα θέλαμε να υπάρξει δηλαδή μια πολιτική συνένεση στα ανώτερα κλιμάκια, ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η συνεργασία και όσο γίνεται μεγαλύ... ευρύτερη επιτόπου. Τώρα βέβαια, όπω και εσείς βλέπουμε την πραγματικότητα και ποια είναι η δυσκολία τη σήμερα ημέρα να ληφθεί μια απόφαση που να δεσμεύει τους 28. Διότι πλέον μπορούμε να μιλάμε για 28 και βλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δομημένη, διαρθρωμένη συνεργασία που δεν έχει ακόμα θεσπιστεί και όλα η συζήτηση σε σχέση με αυτό αφορά το βαθμό ένταξη. Από τη μια μεριά θέλουμε όλοι να συμμετέχουν, να έχουμε κάτι πραγματικά ευρωπαϊκό και κοινό. Ε, αυτό υπάρχει και στη συνθήκη και από την άλλη έχουμε την πραγματικότητα που μας κάνει να τίνουμε να προχωρήσουμε πιο ρεαλιστικά μικρέ ομάδες. Αυτοί που θέλουν και μπορούν να ξεκινήσουν και οι υπόλοιποι στην πορεία να μπουν. Με τον κίνδυνο βέβαια ποτέ να μην μπουν στην συνεργασία. Και έτσι τελικά δεν έχουμε αποφασίσει, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πάντοτε είμαστε ανάμεσα στις δύο αυτές εναλλακτικέ. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι μια προσέγγιση αρκετά ρεαλιστική που θα χρειαστεί να ακολουθηθεί στο Συμβούλιο. Τώρα δεν ξέρω, μισογεμάτο, μισοάδιο το ποτήρι. Στο Συμβούλιο εγώ προσωπικά και αυτό δεν δεσμεύει κανένα, έχω την τάση να ικανοποιούμε με τις μικρές πρακτικές και ρελιστικές συνεργασίες από κάτω προς τα πάνω. Λέω ότι είναι καλύτερο από το τίποτα και αν δεν έχουμε ούτε και αυτό το μήνυμο κινδυνεύουμε να μην έχουμε τίποτα. Ομολογώ ότι ακόμα και ως πεπισμένος Ευρωπαίος ικανοποιούμε με την προσέγγιση την Γαλλογεραβρετανική, την Βελγοολλανδική ή τη Γερμανό-Ολλανδική, λέγοντας ότι είναι καλύτερο και από το τίποτα. Και Έχουμε εδώ λοιπόν μια αποστολή κάπως πιο ψηλή, αν και δεν είναι και πολύ ρεαλιστική, να φτάσουμε δηλαδή σε αποφάσεις που θα δεσμεύουν όσο γίνεται περισσότερες χώρες. Τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω πως πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική τότε. Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι μια σημαντική στιγμή. Θα δώσει μια όθηση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια. Τα κράτη-μέλη ε, ήδη μιλούν για pooling and sharing, smart defense, smart buy. Ξέρουμε τις ανάγκες μας. Σήμερα συζητήσαμε και τις διαδικασίες της Εθνικές Βουλές. Το είπα και προηγουμένως. Θεωρείτε ότι θα γίνει τουλάχιστον έναρξη της συζήτησης ε, των διαδικασιών. Ε, να περάσουμε από τις ε, συναντήσεις τις αποστολές, από τις συναντήσεις τις επιχειρήσεις. Πώς αντιδρούν τα κοινοβούλια και πώς ανταποκρίνονται στις διάφορες κρίσεις του κόσμου. Το Βέλγιο μπορεί να είναι περήφανο για την άμεση αντίδραση που είχε στη Λιβύη. Ενώ σε άλλες χώρες εμάς υπήρξε αρκετή χρονοτριβή. Επίση, την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου έχουμε συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών ότι θα έπρεπε να λάβουμε μέρο, αλλά βλέπουμε ότι οι διαδικασίε είναι πιο χρονοβόρε. Μήπω κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάσουμε και τι διαδικασίε στι εθνικέ ε, βουλέ. Γιατί από την πολιτική βούληση θα ξεκινήσουν όλα. Αυτό απαιτείται. Αλλά η πολιτική βούληση προϋποθέτει και κάποιες διαδικασίες ε, που μερικές φορές ε, εκπορεύονται από τα συντάγματα. Είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από τη συζήτηση, τίποτα δεν θα αλλάξει. Θα δώσω το λόγο στον Έλμαρ Μπρόκ. Γιατί ε, κατάγεται από μια χώρα που δεν λαμβάνονται κοινοβουλευτικές αποφάσεις, τουλάχιστον σε μικρό βαθμό για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Έλμαρ που τα ξέρει αυτά απ' έξω και ανακατοτά. ich Θα äh, äh, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για το θέμα της δομημένης συνεργασίας. Το θέμα είναι πώς ξεκινάει κάτι τέτοιο. Υπάρχει εδώ πέρα διάλογος ε, μεταξύ ε, διαφόρων φορέων, ε, πρέσβεων κτλ. Το θέμα είναι λοιπόν ποιος έχει το δάχτυλο στο σκανδάλι. Γιατί συζητάμε χίλιες μεταβλητές. Και το θέμα είναι τελικά ποιος θα κινηθεί και θα αναλάβει την ηγεσία. Η εμπειρία των τελευταίων μηνών έδειξε πως πρέπει να προχωρήσουμε και γι' αυτό και είπα ότι εκπρόσωπος κάτι θα πρέπει να κάνει παρά το ότι βεβαίως είναι Βρετανίδα και δυσκολεύεται κατόπιν το κόμμα μου ε, επεξεργάστηκε μια ομάδα εργασίας δηλαδή η υποδική μου προεδρία επεξεργάστηκε στη Γερμανία ε, μια πρόταση σύμφωνα με την οποία μετά τις εκλογές ε, θα έχουμε μεγαλύτερη μπλοκή του Κοινοβουλίου και ε, η πρόταση είναι το εξή. Εκεί όπου έχουμε ζητήματα των λεγόμενων enablers, δηλαδή Γερμανοί με στα άβαξ και διάφορα τέτοια, τέτοιες μορφές συνεργασίας, να γίνει μία συζήτηση άπαξ και μετά να μπορούμε να συμμετέχουμε όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές αποστολές αυτομάτως. Και ο τρόπος μετά αλλάξει, να μην λένε συνέχεια άμα τους Γερμανούς δεν γίνεται τίποτα ας πούμε να μπορούν να, μπαίνουν και, να μπαίνει και το γερμανικό πλήρωμα στο αεροπλάνο, στο άβαξ ας πούμε γιατί υπήρχε αυτή η κατάσταση γιατί όπως σας είπα αυτό δεν γίνεται όπως ξέρετε για τις μάχημες θέσεις και αποστολές λόγω συνταγματικών περιορισμών αλλά για τις υπόλοιπες αποστολές ε, πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός για, για να υπάρχει και μία πρακτική λύση και να μην ε, είναι συνεχώς τροχοπέδι η Γερμανία. Μετά τις εκλογές λοιπόν θα γίνει μια συζήτηση και φαντάζομαι πως ε, αυτό το οποίο λένε και άλλα κόμματα είναι πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους. Και οι φιλελεύθεροι νομίζω δεν έχουν κάποιες αντιρρήσεις αρχής. Βεβαίω υπάρχει το ζήτημα του συνταγματικού δικαστηρίου, έτσι. Εκεί πέρα έχουμε το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην πράξη υποθέτω πως το δικό μας το κόμμα δεν θα έχει μεγάλα προβλήματα. Και ελπίζω να προχωρήσουμε και προς το συμφέρον των συμμάχων. Ευχαριστώ. Αυτά σας ευχαριστώ θερμά για την επίσκεψη. και ελπίζω να γίνει πηγή έμπνευση και για άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες. Είμαστε στη διάθεσή σας πάντως. Και κάτι τελευταίο, Στάιντχόβεν είναι έτοιμη η διοίκηση για να σας φιλοξενήσει. Ε, και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αποστολή από την άποψη της προσπάθειας συνένωσης και κοινή χρήση των πόρων. Μάλιστα οικειοθελή συνένωση και κοινή χρήση Πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία αυτή και θα έχουμε όσον που επίσκεψη και θα κάνουμε και μια στάση για να σας ξανασυναντήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για τη φιλοξενία. Ξέρω ότι ήταν έκτακτη αυτή η συνεδρίαση ε, για να προσκαλείτε, έκτακτη συνεδριάση οργανώνεται για να προσκαλείτε και ε, βουλευτές από τις Εθνικές Βουλές. Πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Θα δώσουμε συνέχεια σε τέτοιες ε, συναντήσεις και επαφές και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και σε υπουργικό επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά το pooling and sharing, σίγουρα έχουμε ένα pool αυτό το εκλογικού σώματος και εκεί θα συνεργαστούμε και Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.